So, good morning everybody. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Σήμερα το πρωί έχουμε να συζητήσουμε για την Μύφιτ. Και την προηγούμενη εβδομάδα πήρα κάποιες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις ότι δεν θα εκπλαγούμε και πολύ για αυτά που θα ακούσουμε. Καλωσορίζω λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Στίβεν Μαγιόρ που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ και έχουμε μαζί μας και τον Μάρτι Μαλέρ που είναι ο διευθυντής των χρηματοοικονομικών αγορών. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ως ήθιστε σε αυτόν τον έλεγχο που κάνουμε, το scrutiny slot, μια που πρόκειται για το συνομοθέτη της προηγούμενης χρονιάς, τώρα έχουμε τεχνικές προδιαγραφές 1500 τόσε σελίδες να διαβάσουμε για τη διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότηση τίτλων. Πολύ δουλειά είχαμε να κάνουμε, την κάναμε όμως. Διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε. Περιμένουμε όμως για τι κατεξουσιοδότηση πράξεις και τι εφαρμοστικέ, τα εφαρμοστικά μέτρα να μάθουμε περισσότερα. Όπως πάντα θα αρχίσουμε με την ΕΣΜΑ. Έτσι. Οπότε, παρακαλώ. 10-12 λεπτά ο καθένας. Α, 5 λεπτά. Εντάξει, μαζί 10 λεπτά λοιπόν. Ή 6 ΕΣΜΑ, 4 Επιτροπή, δεν ξέρω, όπως θέλετε. Λοιπόν, έχεις το λόγο, Στίβεν. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκος, 7 λεπτά είχα υπολογίσει, αν συμφωνείτε. Α πούμε ότι είναι ο συμβασμό ανάμεσα στα 5 και τα 10 λεπτά. 7 λεπτά λοιπόν είχα υπολογίσει να μιλήσω. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι. Πολύ χαίρομαι που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή αυτή, την οικονομική, για να σας ενημερώσω για τη ρυθμιστική δουλειά που κάνουμε στην ΕΣΜΑ και να ανταλλάξουμε απόψεις και για το περιεχόμενο της. Όπως γνωρίζετε, δημοσιεύσαμε τέλη Σεπτεμβρίου τις τεχνικές προδιαγραφές για το MIFID 2, για το MAR και για το CSD, το κεντρικό αποθετήριο τίτλο δηλαδή, που μας κόστησε δύο χρόνια. 900 σελίδες κανόνων που λίγο λιγότερο από ό,τι είπε ο πρόεδρο, που φυσικά οδηγούν σε παραπάνω ερωτήσεις που χρειάζονται σε βάθος συζήτηση για το τι μπορούμε να πετύχουμε και τι όχι. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι το προσωπικό της ΕΣΜΑ, παρόλο που εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε πολύ σε βάθος, είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, τι ε, μας κάνει να προβληματιζόμαστε στο τελευταίο αυτό σχέδιο για τις, ε, τις ρυθμίσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι θέλουμε να καταλήξουμε στο πώς θα προσδιορίσουμε κατά πόσο ένα ομόλογο έχει ρευστότητα ή όχι. Ακούσαμε τις ανησυχίες σας την προηγούμενη φορά και εμείς πιστεύουμε ότι με τον τρόπο που προτείνουμε μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς, να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες και να καλύψουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό ομολόγων Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τις υποκείμενες παραμέτρους για να αξιολογηθεί η ρευστότητα μετά την έκδοση ή να αποκλείονται συναλλαγές κάτω από τα 100.000 ευρώ για να καθορίσουμε ποιος μπορεί να υποφεληθεί από εξαιρέσει και από μεταχρονολογημένες δημοσιεύσεις. Έχουμε λοιπόν αρκετές εξηγήσει, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι πιστεύω πως έχουμε ένα σύστημα που πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα αποκλίνοντα συμφέροντα και τον στόχο μας να έχουμε σημαντική διαφάνεια στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων που έτσι θα βελτιωθεί και η λειτουργία τους. Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι το καθεστώς αυτό, το non-equity, της διαφάνειας των non δηλαδή καλύπτει ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών ε, στοιχείων και καλύπτει όλα εκείνα τα στοιχεία που θέλουμε σε λεπτομέρειες. Θα μιλήσω τώρα για τις ε, για τη... τα όρια θέσεων. Θα σας πω ότι λάβαμε υπόψη μας το νούμερο 5 που καλύπτει 35% αντί για το όριο των 10% που μάλλον δεν είναι αρκετά αυστηρό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα συμβάσεις υψηλής ρευστότητας. Αντιλαμβάνομαι ότι παραμένουν κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσο το εύρος αυτό είναι αρκετό ή δεν είναι αρκετό γιατί εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι η ΕΣΜΑ έπρεπε να καθορίσει ένα ευρύ πλαίσιο, μια που το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει έναν τεράστιο αριθμό ε, συμβάσεων, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, που δεν συγκρίνονται με την περίπτωση του Αμερικανικού συστήματος. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω ότι η προσέγγιση της ΕΣΠΑ πρέπει να καταλήξει οι εθνικοί ρυθμιστές να θέτουν αυστηρά όρια όταν αυτά χρειάζονται ή λιγότερο φιλόδοξα όρια όταν αυτό χρειάζεται για να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ρευστότητα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, δοκιμές βοηθητικών δραστηριοτήτων που έχει συζητηθεί πολύ ως θέμα. Θέλω να επαναλάβω ότι η ΕΣΜΑ προσπάθησε να σχεδιάσει τις δοκιμές αυτές προσεκτικά και ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφορικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχουν τεράστιες τεχνικές αδυναμίες όσον αφορά τις δοκιμές για να υπολογιστούν ε, τα κεφάλαια, έχουμε αποφασίσει να δοκιμάσουμε κατά πόσο τα παράγωγα ε, τα εμπορικά αυτά είναι βοηθητικά στις ε, βασικές συναλλαγές. Και αυτό συμμορφούμενοι με το επίπεδο 1. Κάποιοι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν να έχουμε δοκιμές για την κεφαλαϊκή βάση. Αλλά πάλι μερικοί πριν από λίγο καιρό εξέφρασαν ανησυχίε λέγοντα ότι δεν μπορούν να κάνουν τέτοιε κεφαλαϊκέ δοκιμέ, ότι θα κόστιζαν πάρα πολλά χρήματα και δεν θα έδιναν αποτελέσματα συγκρίσιμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πιστεύουμε ότι οι δοκιμέ που έχουμε σχεδιάσει είναι εφικτέ και ευθυγραμμίζονται με του βασικού στόχου των συνομοθετών προκειμένου να μειωθούν οι εξαιρέσει από τον χρηματοοικονομικό κανονισμό, μειώνοντα τα αδιαφανή τμήματα των αγορών και έτσι να μπορέσουν οι μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες να μπορέσουν και αυτοί να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Είμαστε πεπισμένοι ότι μετρήσεις βασιζόμενες στα κεφάλαια θα ήταν ε, τεχνικά μιλώντας αδύναμοι. Θα κόστιζαν πάρα πολλά χρήματα και δεν θα βοηθούσαν στη σύγκληση. Τώρα έρχομαι στις εφαρμοστικές προκλήσεις του έργου μας όσον αφορά τη MIFID. Δεν πρόκειται εδώ να εκπλήξω κανένα σας αν σας πω ότι οι ρυθμιστές και οι επενδυτές δυσκολεύονται πολλές φορές να εφαρμόσουν τους κανόνες. Και επιπλέον υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου το χρονοδιάγραμμα ήδη αποδεικνύεται ανέφικτο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πάρει χρόνο πέρα από το 2016 πριν να έχουμε ένα τελικό κείμενο για τις ρυθμίσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Μπορούν λοιπόν όλα αυτά να ξεκινήσουν μόνο όταν έχουμε πλήρω τι λεπτομέρειε τη RTS, τη ρύθμιση δηλαδή τεχνικών προδιαγραφών και μετά θα χρειαστεί άλλο ένα χρόνο. Συνεπώ, θέτουμε το θέμα αυτό του χρονοδιαγράμματο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέμε ότι κάποια συστήματα πληροφορική δεν θα είναι έτοιμα πριν από το 2017 και αναφίβολα αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίε για την εκτέλεση κάποιων στοιχείων τη MIFID 2. Επιπλέον, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε συζητήσει κατά πόσο η αβεβαιότητα αυτή χρειάζεται μια νομοθετική απάντηση για να δούμε τι θα γίνει τελικά με τη MIFID 2 για να πετύχουμε την διαφάνεια στις συναλλαγές και την αναφορά των όσων συμβαίνουν στις συναλλαγές αυτές. Η αναφορά λοιπόν των ε, συναλλαγών απαιτεί να δημιουργηθούν νέα πληροφοριακά συστήματα από την αρχή και στις διάφορες πλατφόρμες διαπραγματεύσεων και είναι δύσκολο να καταφέρουν όλοι αυτοί να είναι έτοιμοι για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συγκρισιμότητα. Επιπλέον, οι επενδυτικές επιχειρήσεις και οι πλατφόρμες συναλλαγών χρειάζονται σημεία αναφοράς και πρέπει όλα αυτά να γίνουν από την αρχή. Για να έχουμε λοιπόν τέτοια πληροφοριακή υποδομή μας χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουμε να δημοσιεύουμε έναν ενίο κατάλογο συναλλαγών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όρια από τα οποία απαιτείται η διαφάνεια. Όλα αυτά τα σχέδια είναι τεράστια και περίπλοκα. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στην ΜΥΦΙΔ 1, όπου απαιτήθηκαν τρία χρόνια για την εφαρμογή της. Αυτά τα σχέδια εφαρμογής καταλαβαίνετε ότι μας δείχνει το εύρος των δραστηριοτήτων που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σωστός συντονισμός από την έγκριση της αρτιές, την μεταφορά της εθνικής νομοθεσίας, της κατεξουσιοδότηση πράξης και την πληροφοριακή υποδομή και τη δημιουργία της. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει το Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Στίβεν ήταν πολύ περιστατωμένο και γι' αυτό εγώ μπορώ να είμαι πιο σύντομο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Φέμπερν, ε, ε, την κυρία Σουίνμπορν, τον κύριο την την κύριο Φανόβερνάιζεν, τον κύριο Κέγκολτ και τον κύριο Ντεμάση για την υποστήριξή του στη διάρκεια ολόκληρη τη ε, διαδικασία του ΜΥΦΙΤ. Βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε αυτή τη συζήτηση για τα πιο κύρια θέματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ΕΣΜΑ που μας έδωσε αυτές τις πολύ περίπλοκες τεχνικές προδιαγραφές. Είναι ένα μέγα επίτευγμα. Είχαμε πολύ αυστηρές προθεσμίες. Καλωσορίζουμε το πακέτο που ε, υπευλήθη και νομίζω ότι αυτό στρώνει το δρόμο για να έχουμε ένα ενιαίο κώδικα ε, για τις ε, επενδυτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Ο Στίβεν επίσης παρουσίασε τα κεντρικά ζητήματα που θα απαιτήσουν πολύ μεγάλη προσοχή στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της διαφάνειας, την επέκταση των απαιτήσεων διαφάνειας σε ένα μέγα ε, φάσμα άλλων τάξεων ενεργητικού, πράγμα που είναι μια μεγάλη πρόκληση και η ΕΣΜΑ χρειάστηκε να αναπτύξει μια τελείως νέα μεθοδολογία ώστε να φωτίσει τον σχηματισμό της τιμολόγησης στον τομέα στις αγορές των ομολόγων και των παραγόγων. Οπότε βλέπουμε το τελικά σταθμισμένο αποτέλεσμα της εργασίας της ΕΣΜΑ και το εξετάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Στη συνέχεια το θέμα των μη χρηματοπιστωτικών εταιριών που εμπορεύονται ε, παράγωγα αγαθών και εδώ η ΕΣΜΑ χρειάστηκε να βρει μια ανισορροπία ανάμεσα στην κάλυψη των μεγάλων κερδοσκοπικών εμπόρων παραγόγων χωρίς όμως να σταματήσουν θεμητές, χωρίς να υποβάλουν μάλλον θεμητές δραστηριότητες ε, hedging στην ε, οδηγία MIFID. Και τρίτον, Έχουμε τα όρια θέσεων που γνωρίζουμε πως ήταν δύσκολο για την ΕΣΦΑ να σταθμίσει αυτά τα όρια με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει την μεγάλη ποικιλία συμβάσεων που θα καλύπτονται από το καθεστώς ορίων θέσεων που αποφάσισε ο νομοθέτης. Και αυτό είναι άλλο ένα θέμα λοιπόν το οποίο ε, ε, τραβά την προσοχή μας. Για όλα αυτά τα θέματα αλλά και για όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάποια θέση από πλευρά της Κομισιόν ακόμη. Αξιολογούμε την εργασία από τεχνικής και νομικής άποψης. Παράλληλα εργαζόμαστε σκληρά επί των τριών ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων που ελπίζουμε να υιοθετήσουμε σύντομα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε τις κατεξοδότητες συμπράξεις και τα τεχνικά, τις τεχνικές προδιαγραφές να εγκριθούν έτοιμα ώστε να εγκριθούν όσο γίνεται πιο σύντομα το 2016 και να αρχίσουν να εφαρμόζονται και το 2000, μάλλον να δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα μέσα στο 2016. Τίποτα δεν θα, μας πρέπει, δεν θα πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό το στόχο. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε ότι η MIFID αποτελεί ένα, μια βασική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι αγορές, απαιτεί μεγάλες προσπάθειες για τη συλλογή και την ε, επεξεργασία των εμπορικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό είναι κάτι για το οποίο η ΕΣΜΑ, οι εθνικοί ρυθμιστές αλλά και ο ο κλάδος ο εμπορικός χρειάζεται χρόνο για να, το, για προσαρμοστούν σε αυτό. Ο Στίβον ανεφέρθηκε στην ανάγκη μάλλον κάποιες καθυστέρησεις στην εφαρμογή του πλαισίου της ΜΥΦΕΝΤΟ ώστε να υπάρξει ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του πακέτου. Όντως ε, λάβαμε ε, σχετικό σημείο από την ΕΣΜΑ ως προς αυτό και αυτό το αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Η ε, αρχική μας ε, τεχνική φύσης θέση είναι ότι όντως χρειάζεται μια καθυστέρηση. Εάν θέλουμε να έχουμε ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή, θα χρειαστεί να αποφασίσουμε και να συζητήσουμε μαζί μεταξύ μας ποιο θα είναι το φάσμα και η διάρκεια αυτής της καθυστέρησης. Και πάλι η πρώτη προκαταρκτική προκαταρτική μας θέση είναι ότι ίσως το απλούστερο και νομικός βάσιμο θα ήταν να καθυστερήσει κατά ένα έτος ολόκληρο το πακέτο. Αλλά είμαστε έτοιμοι και διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί σας και με το Συμβούλιο άλλες επιλογές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα, ως πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και μετά στους κοιόδης. Είμαι και εισηγητή βέβαια εγώ ίδιο, οπότε θα τα πω στα γερμανικά και είναι δύσκολα και περίπλοκα τα θέματα, αλλά θα τα πω και εγώ στα γερμανικά. Σε ευχαριστώ πρώτα που ερχόμεθα πάλι να συζητήσουμε για την οδηγία MIFID και ομολογώ ότι εκπλήσωμαι διεξάγεται τέτοια συζήτηση με ΕΣΜΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τέτοιο χρονικό σημείο. Είχα γράψει στον ε, Επίτροπο για να ρωτήσω πότε θα υποβάλει τις εφαρμοστικές και εκτελεστικές πράξεις. Είπε φθινόπορο 2015. Το φθινόπορο πηγαίνει μέχρι... Ε, τελειώνει σε λίγο. Τώρα λέει αρχές 2016. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωσή του και μετά από αυτό χρειάστηκε περίπου 9 μήνες το Συμβουλίο μέχρι ότου είναι έτοιμο για να συζητήσει μαζί μας. Η Κομισιόν, και το λέω καθαρά, ήδη απέτρεψε μια πρώτη συμφωνία το 2013. Από τότε γνωρίζουμε βέβαια τα κείμενα. Τον Απρίλιο του 2014 ενέκρινε τα κείμενα το Κοινοβούλιο, το ΔΕ Συμβούλιο τα ενέκρινε λίγο μετά. Και μέχρι τέλους μιλούσαμε διαρκώς και για το χρονοδιάγραμμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ΕΣΜΑ. Βεβαίω είναι το θέμα περίπλοκο, το γνωρίζω και ήταν εξ αρχής σαφές και όλοι γνωρίζαμε η δουλειά σημαίνει το θέμα αυτό. Μπορώ να σας επαναλάβω διάφορες συνομιλίες που διεξήγαγα και ε, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Έτρεχα από πίσω σας και προσπαθούσα να διευκρινίσω τα πράγματα για λογαριασμό του κοινοβολίου στην στον τελευταίο τριμερή διάλογο τον Ιανουάριο μιλήσαμε για τις ημερομηνίες. Εγώ βεβαίω ήμουν απολύτω ανοιχτό να μιλήσω μαζί σας σοβαρά για τις ημερομηνίε. Με βεβαιώσατε ότι τα πράγματα προχωρούν. Με βεβαίωσαν ότι μέχρι τα μέσα του φετινού χρόνου θα είχαμε τα κείμενα από την Κομισιόν. Και μόλις προλίγου έλαβα επιστολή από τον Επίτροπο ότι θα έλθουν τον, το, το φθινόπωρο του 2015. Τι να σας πω, δεν μας έχετε προκαλέσει μεγάλη χαρά με όλα αυτά, με τις αναβολές επί αναβολών, της εφαρμογής του θεμελιώδους ε, λίθου, του θεμέλιου καλύτερα λίθου, για την, ε, ε, τις επενδυτικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιλούμε για τις υποχρεώσεις που έλαβαν το 2000, ανέλαβαν το 2009 οι χώρες μέλη στα πλαίσια του G20. Και είμαστε το τμήμα εκείνο του κόσμου το οποίο χρειάστηκε και περισσότερο χρόνο για να οργανωθεί για τα πράγματα αυτά. Βεβαίω η MIFID 2 είναι πλέον περίπλοκη από την MIFID 1, αλλά βεβαίω συζήτησα και με του σκιώδει συγητές εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών. Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε το δυνατόν συντομότερο ε, συζήτηση με τον Επίτροπο και με τις ε, αρχές της ε, Κομισιόν και να δούμε ποια πράγματα μπορούμε ενδεχομένω να εφαρμόσουμε ταχύτερα θα έρθω σε ορισμένα θέματα και το ερώτημα που τίθεται πάντοτε είναι αν έχουμε επαρκή δεδομένα. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα και είναι και τα διάφορα θέματα της εφαρμογής του ΕΜΙΡ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε σύντομα και σύμφωνα με το πρόγραμμά μας την επόμενη εβδομάδα ήδη να διεξαγάγουμε τη συζήτηση αυτή για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες, ιδίω για τον φύρ, τον κανονισμό, δηλαδή ο οποίος ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται εν μέρει ορισμένα τμήματα του Σιουνίδη και να δούμε ποια άλλα μπορούν να τεθούν ταχύτερα σε ίσχυ. Και το ότι πρέπει τώρα να αναβάλουμε για άλλο ένα χρόνο το τμήμα περί που είναι ο πυρήνας της ε, νομοθεσίας MIFID για να γίνουν πιο διαφανείς οι αγορές και πιο σταθερές. Τώρα αυτή η αναβολή εμένα με ανισχύει πολύ, το λέω καθαρά. Έχω πάντως ορισμένα θέματα τώρα, τα οποία ε, επίσης με ανησυχούν. Η, τα position limits από την επιστολή που στείλαμε στην ΕΣΜΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφές ότι τα όρια θέσεων είναι ε, θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι είναι και περίπλοκο. Αν θέλει κανείς να ασχοληθεί με όλα τα είδη παραγόγων, ε, στην ουσία ψάχνει λίγο στα τυφλά. Υπάρχει όμως μια καθορισμένη τιμή, 25% και από εκεί και πέρα είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω μπορούν να απεικονιστούν όλες οι αγορές. Εγώ όμως αυτό το αμφισβητώ και εκπλήσωμαι που τα διάφορα όργανα το έχουν δεχτεί αυτό το πράγμα. Γιατί για πολλοί ασταθείς αγορές είναι πολύ υψηλές οι τιμές αυτές. Σε μια πολύ ασταθή αγορά ήδη και το 5% των positions είναι υπερβολικά πολύ. Για πιο σταθερές αγορές. Παράδειγμα, το LNG, το ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπου έρχονται λίγα από τα προϊόντα αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά, καράβι-καράβι, και υπάρχει μικρή αγορά. Ήδη εκεί το 35% είναι υπερβολικά μικρό. Θα καταρρίψει η αγορά αυτά με τις προτάσεις που κάνετε. Δηλαδή, η απάντηση που δίνεται αναφέρεται μοναχά σε ένα μικρό τμήμα των παραγόγων. Για το μέγα όγκο των ε, εμπορευμάτων δεν απαντάτε στο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγιστεί το θέμα διαφορετικά. Όχι γραμμικά, αλλά τουλάχιστον με δύο διαστάσεις και με, με ένα μάτριξ για να μπορούν να προβλέπονται διάφορε παραλλαγέ. Για εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά που λέτε, οι προτάσεις σα για τα position limits εξακολουθούν να μην είναι αποδεκτέ. Διότι ιδίω στον τομέα των τροφίμων δεν απαγορεύει αυτά που θέλουμε να απαγορεύσουμε γιατί είναι υπερβολικά υψηλέ οι τιμέ. Και για ειδικά προϊόντα και σε ασταθεί αγορέ θα οδηγηθούμε τελικά στο να ε, εξαφανιστούν οι αγορε αυτέ. Δεν μπορεί όμω κάτι τέτοιο να είναι ο σκοπό να αλλάξουν δηλαδή οι αγορές να είναι τέτοιο πράγμα ο σκοπός των ε, προτύπων αυτών. Εδώ λοιπόν έχουμε δημιουργήσει εξαίρεση στην νομοθεσία, την προτείνουμε εμείς δηλαδή, επίτηδες η ΕΣΜΑ προβλέπει να βρεθεί λύση με ε, μια δοκιμασία σε δύο φάσεις, market και main market. Εγώ έχω πάλι εδώ ορισμένε επιφυλάξει. Η επιστολή μας αναφερθήκαμε μοναχά στις τιμές κατοφλίων, σε και τιμές, όχι στο ίδιο το σύστημα. Εκεί χρειάζεται περισσότερη επιχειρηματολογία γιατί γίνεται δηλαδή αυτή η συστημική αλλαγή. Και για το μέλλον δεν έχουν υποβληθεί αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία για τις αγορές. Δεν μπορεί λοιπόν καν να ελεγχθεί το τμήμα της αγοράς, το ποσοστό δηλαδή της αγοράς και πώς θα υποβάλλετε το δυνατόν συντομότερο τα δεδομένα. Λέτε εδώ, άμα τη θέση σε ισχύ. Πώς θα γίνει αυτό όμως. Μετά, το ζήτημα το, τους κανόνες ρευστότητας. Είπαμε, μια προσέγγιση αναμέσων, instrument by instrument. Για τους πρώτους έξι μήνες μετά από νέα, ε, νέο δάνειο, λέτε εδώ, classes of financial instruments, να ρυθμιστούν αυτά. Εγώ θέλω μια εξήγηση να μου δώσετε εδώ, γιατί δηλαδή ακολουθεί το δρόμο αυτό. Επίσης, εν ώψη των σχετικά χαμηλών οριακών τιμών για τους εμπορικούς όγκους, βλέπω ορισμένα να ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως ρευστά εν τέλει, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είναι. Τα πρώτα, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό. Μήπως λοιπόν τίθεται το ερώτημα, είναι οι οριακές αυτές τιμές υπερβολικά χαμηλές. Και για τα SSTI waiver για όρια τιμών κάτω των 100.000 ευρώ. Αλλιώς οι εμπορικές, ε, ο εμπορικός όγκος δεν θα είναι επαρκής και ενδέχεται να ε, παρισφρήσουν σφάλματα. Στα τελευταία σχέδια, στο RTS2, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα αγορά, στην πρωτογενή αγορά. Και τελικώ καθίσταται άχρηστο αυτό λόγω έλλειψη διαφάνεια. Επομένω εδώ η διατύπωση είναι λιγότερο ακριβή από την παλιά και εδώ χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Για το θέμα τη πρόσβαση. Η ΕΣΜΑ δέχεται τι πρώτε προτάσει του Κοινοβουλίου. Ωραία, θετικό αυτό. Στο άρθρο 12, στο RTS 15, λέει ταυτόσιμη αντιμετώπιση όλων των συμβάσεων, δηλαδή μη διακριτική μεταχείριση όλων των ε, συμβάσεων. Αυτό θα ήταν ωστόσο η δεύτερη αυτή διατύπωση, θα ήταν η πλησιέστερη σε αυτό που επιθυμεί ο νομοθέτης. Και τώρα για το Transaction Reporting στο RTS 23 και 24, η ΕΣΜΑ αναφέρεται στους αριθμούς ταυτοποιήσεως τους διεθνείς αριθμούς ταυτοποίησεως, ίσο 1 λοιπά Και αυτά ρυθμίζουν όλα τα μέσα τα οποία ε, χρησιμοποιούν οι αγορές. Εδώ υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα παράγωγα OTC. Γιατί επέλεξε η ΕΣΜΑ αυτά τα πρότυπα και απέριψε την ιδέα να χρησιμοποιήσει άλλους αριθμούς ταυτοποίησεων. Θα παραμείνω σε αυτά το πιο κρίσιμο από όλα για μας είναι το χρονοδιάγραμμα. Τώρα υπάρχει, είναι εδώ παρούσα και η Ανελίση Ντότς από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φέρμπερ, για τη σκληρή δουλειά που κάνει. Πραγματικά το εκτιμά όλος ιδιαίτερος και είμαι και ευγνώμων για την υπομονή σας όταν πριν από δύο εβδομάδες είχα και εγώ γρήπη και τα φορτωθήκατε εσεί. Ευχαριστώ πολύ και τους προσκεκλημένους μα που ήρθαν εδώ για τον έλεγχο αυτό που γίνεται βέβαια σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι χάρη στην ε, ηγετική θέση του κύριου Φέρμπερκ καταφέραμε και εμείς να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να περιοριστώ στις παρατηρήσεις μου και να επικεντρωθώ κυρίως σε δύο θέματα. Πρώτον την αναβολή και δεύτερον στα όρια θέσεων. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την αναβολή. Εννοείται, πρόκειται και κάτι καινούριο, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που συνδέονται με την προσέγγιση που προτείνεται και πρέπει να δώσουν περισσότερη σημασία στην ίδια την ε, ουσία της ρύθμισης. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την επιθυμία των εισηγητών να έχουν συνάντηση με όλες τις πλευρές και να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσει αυτή η αναβολή. Είναι ζωτική σημασία. Λοιπόν, η πρώτη μου ανησυχία είναι ότι οι διαδόσεις για την αναβολή κυκλοφορούν εδώ και καιρό, το ξέρουν οι συνάδελφοι. Και κάποιοι βλέπαν την αναβολή σαν μια ευκαιρία να ξανανοίξουν κάποιοι από τους δύσκολους συμβιβασμούς τους οποίους καταλήξαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα διάφορα, διάφορες άλλες πλευρές εδώ και μήνες. Πολλά στοιχεία της ε, MIFID 2 προφανώς και είναι επίμαχα, αλλά η αναβολή αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για τα λόμπι, στο οποίο εδώ και μήνες βέβαια μου προσεγγίζουν, για να ξανανοίξουν αυτά τα ζητήματα και να το δουν σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να υποβληθούν νέες τροπολογίες και να γίνουν και άλλες αλλαγές. Αν υπάρχει αναβολή, αυτή θα πρέπει να έχει να κάνει μόνο με τα στοιχεία τα οποία είναι πιο προβληματικά και όπου υπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές προκλήσεις και όχι για ολόκληρο το εύρος της ρύθμισης. Δεύτερον, όσον αφορά το πόσο θα κρατήσει αυτή η αναβολή. Και πάλι ευχαριστώ τους συζητητές που είπαν ότι και αυτό πρέπει να συζητηθεί με λεπτομέρειες. Όντως, αν είναι πολύ μεγάλη η περίοδος αυτή η αναβολής, τότε καταλαβαίνετε ότι θα χάσουμε το ρυθμό μας. Οι συνάδελφοι θα νιώσουν, α, την έχουμε αυτή την αναβολή που τη θέλαμε, εντάξει, τώρα μπορούμε να ευσυχαστούμε» και ας περιμένουμε για μήνες. Οπότε μετά από μήνες θα καταλήξουμε να ξανασυζητάμε τα ίδια προβλήματα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δεδομένου των προβλημάτων που οδήγησαν στην αναθεώρηση της MIFID, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο συγητής, να δούμε τις προτεραιότητές μας. Πολύ σύντομα τώρα. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα των position limits, των ορίων θέσεων και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να συζητήσω γιατί όπως είπατε και εσείς είναι ζωτική σημασία για το Κοινοβούλιο και για την δικιά μου την πολιτική ομάδα. Όπως θα θυμόσαστε όλοι, πολλές φορές μέχρι τώρα έχω πει ότι προσωπικά πιστεύω ότι η βασική γραμμή πρέπει να... Ε, το 25% μάλλον είναι πάρα πολύ ψηλό Δεδομένου ότι η ΕΣΜΑ έχει κάνει αλλαγές για το καθεστώς όπως είπαμε και σήμερα από το 10 στο 40 στο 5,35%, το μήνυμα που στέλνουμε στις αρχές ανταγωνισμού είναι ότι με το 25% μπορούν να θέσουν τα όρια για, τα, για τις συμβάσεις ρευστότητας ψηλά. Έχω ακούσει τις θέσεις της ΕΣΜΑ τις επανέλαβε και σήμερα, πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τις εθνικές αρχές για να θέτουν τα όρια αυτά. Αλλά συγχρόνως έχουμε παραδείγματα από τη Γαλλία για παράδειγμα όπου με το Martic που είναι τα πιο βασικά ενεργειακά συμβόλαια στην Ευρώπη που ήταν 35%. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τωρινές αναλογίες. Και ξέροντας ότι το 25% το ανώτατο όριο συχνά στις Ηνωμένε Πολιτείε και όχι το όριο από το οποίο ξεκινάει, πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι σοσιαλιστές θέλουν μια βασική γραμμή 25% ή χαμηλότερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεισαγάγει κριτήρια για την ε, ρευστότητα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάνω σε αυτό. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το βασικό ζήτημα είναι η αναβολή. Καλό είναι που έχει εμπλακεί το Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών μας οργάνων, τις αποφάσεις αυτές να τις παίρνουμε σωστά και προσβλέπω σε συζητήσεις στη διαπραγματευτική ομάδα και με την Επιτροπή. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Και Σίλμπρουκ από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, και όλους όσους εργάστηκαν πάνω σε αυτό το θέμα για τα τεχνικές προδιαγραφές. Άρα λοιπόν μια ιδέα, μια πρόταση για πιθανή καθυστέρηση δεν κατεβαίνει και πολύ εύκολα, δεν καταπίνεται και πολύ εύκολα. Ε, ξέραμε βέβαια ότι η Μίφιντα από την αρχή δεν θα ήταν πολύ εύκολη και γι' αυτό θέλω να τονίσω ένα-δυο στοιχεία στο θέμα των τεχνικών τεχνικών προδιαγραφών ε, που, δεν, ε, που θέλω να αποσαφινιστούν και κάτι θα πω για την καθυστέρηση στο τέλος. Δεν είναι εντυπωσιακό λοιπόν πως αυτό το, το θέμα εξακολουθεί να είναι ε, η το καθεστώ διαφάνειας για τα non-equity. Το έχω πει 100.000 φορέ όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως δεν έχει νόημα να έχουμε ένα πρόγραμμα για ένωση των κεφαλαγορών εφόσον οι εταιρείε δεν θέλουν ε, και οι διαχειριστές δεν θέλουν να ορίσουν τι είναι ρευστότητα. Το πρώτο καθήκον ήταν το να οριστεί μια ρευστή αγορά έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής αγοραπολισία και δεν νομίζω πως το δυο φορές την ημέρα ορίζει την αγορά ρευστότητας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κατά πόσο Δέκα φορέ την ημέρα που χρησιμοποιούμε για άλλα παράγωγα ή για άλλα μέσα θα ήταν καταλληλότερο ως μήνυμο στάνταρ για την εμπορία non-equity. Επίσης θα ήθελα να δω, ε, όπως και ο εισηγητής, πιο λογικό όριο για το SSTR ή αν όχι για όλα τα μέσα non-equity έτσι ώστε να μην αποθαρρυνθεί η δημιουργία αγοράς. Ωστόσο αυτό δεν υπάρχει σε αυτήν την πρόταση. Θα ήθελα ωστόσο να πω δύο πράγματα ε, μετά από τη δημοσίευση του ΕΣΜΑ, τα ανέφερα και στη Βρετανία, αλλά θέλω να ακούσω εδώ πώς θα απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις που αναφέρθηκαν στο τέλος αυτής της διαδικασίας τον περασμένο μήνα και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πληρέστερες απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα εδώ υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου ε, καθένα θεωρούσε ότι η ανάπτυξη αγοράς ε, ΡΣΜΗ ήταν ε, μια επέκταση της αγοράς. Το ITS 19 φαίνεται να προσθέτεται κάποιες κάποιες απαιτήσει, ενώ υποτίθεται ότι το απλοποιούμε το σύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν τα προσθέτεται εδώ. έπειτα, οι αναφορές για την και μου είπαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι ότι αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και 36.000 ε, σημεία ως στοιχεία. Δεν το πιστεύω ότι θα είναι τόσο μεγάλο. Όμως εσείς μπορείτε, έχετε μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε ποια τάξη μεγέθους συζητάμε. Έπειτα, οι απαιτήσει αναφορά για την εκτέλεση όπω έχουν σχεδιαστεί είναι αυτό συμβατό με τη διαφάνεια όπω προτείνονται για το πρότυπο RT, ε, δηλαδή για τα τεχνικά, τι τεχνικέ προδιαγραφέ. Και έπειτα, οι κώδικε που έχουν θεσπιστεί στον τομέα των χρεογράφων, securities, πώ θα εντοπιστούν και πώ θα χρησιμοποιηθούν για όλα ε, τα υπόλοιπα μέσα, για να μπορέσουμε να τα εντοπίζουμε δηλαδή. Επίση θέλω να καταλάβω με ποιο τρόπο θα έχουμε ερωταπαντήσεις και επαφή με την ΕΣΜΑ. Να έχουμε δηλαδή μια διαφανή διαδικασία σε σχέση με το Κοινοβούλιο, έλεγχο αν αυτό είναι απαραίτητο, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαδικασία ερωταπαντήσεων. Επίσης να αναφερθώ στο θέμα που εσείς αναφέρατε σε σχέση με τα πακέτα προϊόντων ε, και τις ε, προδιαγραφές διαφάνειας. Πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, σας έχω ήδη πει ότι το να καθυστερήσουμε όλο αυτό το πακέτο για ένα χρόνο, κατά τη γνώμη μου, είναι δυσάρεστο. Πάντως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε η αναφορά των στοιχείων, εάν υπάρξει ε, καθυστέρηση, να ξεκινήσει νωρίτερα, ώστε να υπάρχει μια βελτίωση της στάθμισης των κατοφλίων, των καθεστώτων, αλλά και των ορισμών σε, όπως, σε τομείς, όπως η ρευστότητα των ε, μέσων non-equity. Αυτά να γίνουν δηλαδή πριν ε, από την συνολική εφαρμογή του πακέτου, αν αυτή καθυστερήσει. Εγώ θα ήθελα να γίνουν όλα σωστά, ακόμα και αν μας πάρει παραπάνω χρόνο. Το καταλαβαίνω ότι και εσείς αυτό ζητάτε, όμως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μια καθυστέρηση θα σημάνει καλύτερα στοιχεία για οποιαδήποτε στάθμιση. Επίσης, οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ελέγχους των διαφόρων μοντέλων ε, όσον αφορά τα καθεστώτα διαφάνειας που έχουν προταθεί. Αποτελεσματικά, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί η, ο παραπάνω χρόνος, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως όταν όντως εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα θα είναι δικαιότερο. Η εφαρμογή του MIFID τέλος θα πρέπει να οδηγήσει σε δίκες και αποδοτικές κεφαλαγορές για ολόκληρη την Ένωση. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σταθερά μέσω της αυξανόμενης διαφάνειας και της αποκάλυψης των στοιχείων. Δεν θέλουμε όμως να καταστρέψουμε την αγορά ομολόγων μας. Οτιδήποτε λοιπόν βελτιώσει την εφαρμογή ώστε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά για να εγκρίνω καθυστέρηση ολόκληρου του πακέτου θα πρέπει να είμαι πεπισμένη ότι έχουμε ε, στόχο την καλύτερη εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Και, και τώρα ο Φάμπιο Ντεμάση από την Γκουε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους όσους έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Καταρχήν θέλω να υποβάλει την ερώτηση προς την ΕΣΜΑ. Από ό,τι γνωρίζετε ότι υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής Γιατί και ο εισηγητής μας ε, ε, έμεινε έκπληκτος. Κατανοώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όταν ε, είναι μια τόσο μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια και περίπλοκη, αλλά πάντως δεν πρέπει αυτό να είναι δικαιολογία ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να καθυστερήσουν τη δική τους εργασία. Αυτό είναι άλλο ε, θέμα. Η συλλογή των στοιχείων θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Δεν είναι το πρόβλημα της ε, τεχνολογικό, είναι θέμα ε, ρυθμιστικό. Σαφώς Δε υπάρχει δυσαρέσκεια με τα αποτελέσματα της εργασίας της ΕΣΜΑ σε διάφορες ε, ε, περιπτώσεις. Εγώ πιστεύω πως αυτό το επίπεδο RTS δεν αντιστοιχεί στη συμβιβαστική του πρώτου επίπεδου, ούτε θα επιτυχάνεται κατά τη γνώμη μου ο στόχος της MIFID. Η Κομισιόν ε, θέλει να τροποποιήσει το RTS έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην χρειάζεται να το αλλάξει και πάλι. Οι αλλαγές που έκανα η ΕΣΜΑ από το 10 στο στους 35 είναι βελτίωση, αλλά είναι λιγοστή και μη επαρκής. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω τα όσα είπε και αναλύς. Δεν είμαι πεπισμένος. ξακολουθώ να μην έχω πιστεί από κάποιο τεχνικό επιχείρημα για το ότι η αγορά στη ΣΥΠΑ είναι τόσο διαφορετική και άρα τα δικά μας όρια θέσεις θα πρέπει να είναι τόσο χαλαρά. Συμφωνώ ότι θέλουμε διαφορετικά όρια για τις διάφορες αγορές. Αυτό εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να είμαστε τόσο πολύ εκτός των όσων βλέπουμε να γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Τώρα, η βασική θέση ότι το μύφι πρέπει να είναι χαμηλότερο από το 25% αλλά τα όρια ε, σύλληψης θα πρέπει να είναι σημαντικά ψηλότερα. Αν επιλέξουμε λοιπόν αυτήν, αυτόν τον ορισμό ε, θα πρέπει τα όρια να είναι ε, ψηλότερα. Έπειτα, ο ορισμός και το κατόφλι που ορίζεται για το δικημή βοηθητικών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά ψηλός. Αυτή είναι τα σχόλιά μου και για να μπορέσουμε να έχουμε τη διαφάνεια αλλά και να μπορούμε, μπορεί και ο κλάδος αυτός να προβλέψει, πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να μην συνεχίσουμε αυτό το είδος του ping-pong, γιατί όσο το συνεχίζουμε τόσο περισσότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε όπως αυτά που μας εξηγήσατε σήμερα, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο ε, για το πώς θα σχεδιαστεί η μελλοντική ε, αυτή διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ Φάμπιο. Σας ευχαριστώ Φάμπιο. Ο Φίλιπ Λάμπερτ των Πράσινων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα όσα εξηγήσατε στην εισαγωγική σας ε, τοποθέτηση. Έχετε απόλυτα δίκιο, Πρόεδρε. Κύριε Μαϊόρ, εάν εργαζόμουν στην χρηματοπιστωτική, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, μπορεί να μην το δεχόμουν βέβαια ανοιχτά γιατί θα ήταν υπερβολικά προφανέ, Θα ήμουν όμω πολύ χαρούμενο με αυτά που κάνετε, διότι βέβαια οι ομάδε σα έχουν δουλέψει πολύ για να φτιάξουν τα RTS, αλλά όπω είπε ο Φάμπιο πριν, αποκλίνεται σημαντικά από τις προθέσεις του νομοθέτου. Και σας υπενθυμίζω ότι εσείς δεν είστε νομοθέτης. Βοηθάτε τον νομοθέτη, αλλά δεν είστε νομοθέτης. Ακούγοντας δε ότι ζητάτε και άλλη αναβολή, τότε εγώ ως χρηματοπιστωτικός, ως, ε, ε, ε, ως εργαζόμενος στον κλάδο αυτό, θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχής, διότι θα μου δίνατε μια ανάσα ακόμα. Εγώ νομίζω ωστόσο ότι πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί να κερδίσουν πραγματικά το ψωμί τους. Η μύφη είναι δύσκολη υπόθεση, ναι. Χρειάζεται πολύ και σκληρή δουλειά, ναι. Ας αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Συνεχίστε λοιπόν την πίεση, μη τους αφήνετε να αναπνεύσουν. Εν τέλει πάντως δεν έχω δουλέψει ποτέ στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Είμαι νομοθέτης και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνετε. Καθόλου δεν το διασκεδάζω. Διότι πρώτον, όταν σας γράφουμε και υποβάλλουμε μια σειρά ετοιμάτων για να σας ε, εξηγήσουμε προς τα που θέλουμε να κινηθούν τα RTS, πρέπει εσείς να υπακούσετε στην, ε, ε, στις επιθυμίες του νόμοθέτου. Εμείς θεωρούμε ότι έχετε απολύτως αγνοήσει τις επιστολές που σας έχουμε αποστείλει και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στα σχέδια αρτίες. Γιατί πρώτον ε, δέχεστε το open interest αντί για το deliverable supply ενώ το open interest μπορεί να φουσκωθεί όποιος θέλει κανένας. Για να αποφύγει κανείς αυτό το position limit πολύ αρκεί για να λύσει το πρόβλημά του να φουσκώσει Αυτό που λέμε. Και όταν μιλούμε για position limits, ε, εμείς θέλουμε να ε, λαμβάνετε υπόψη η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θα είναι το μέτρο μας, το benchmark. Δεύτερο, ορίζεται όταν μετράτε τα position limits, είναι ένα μέτρο κάποιου πράγματος και το κάνετε τόσο εξειδικευμένο που πάλι εδώ δίνεται τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τα position limits, φτιάχνοντας κάτι που θα είναι πάρα πολύ κοντά στο μέτρο του position limits, που δεν θα ε, μετράει όμως στον παρονομαστή. Τα κάνετε λοιπόν τόσο εξειδικευμένα, που μπορούν να, μπορεί να υπάρξει τελικά σύγχυση ανάμεσα στις συμβάσεις και ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγουν από το position limit είναι να φτιάξετε ένα contract, μια σύμβαση, σε ένα συμβόλαιο σε, κάποια, σε κάποιον άλλο τόπο, σε κάποιο άλλο venue. Πάλι λοιπόν διευκολύνεται αυτούς που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Πολύ καλά τα είπε ο Μάρκος Φέρμπερ όταν αποφασίζεται ότι το benchmark το όριο θα πρέπει να είναι 25% όταν ρευστή αγορά και ακόμα και το 5% είναι υπερβολικό. Αν χρησιμοποιήσω παρόμοια, αν συγκρίσιμα νούμερα με τις ΗΠΑ και αν χρησιμοποιήσετε τα deliverable supply, εκεί το όριο είναι 2,5, ούτε καν 5%. Έχετε μετακινηθεί κάπως βέβαια, αλλά έχοντας υπόψη και τα, τις, και τα βασικά μετρικά, το basic metric, και τον ορισμό του τι σημαίνει σύμβαση, αποδεικνύεται τελικά ότι δεν θα υπάρχουν καν τα position limit. Και στο κείμενο επίπεδο 1 λέμε ζητούμε η μεθοδολογία των υπολογισμών να λαμβάνει υπόψη και την αστάθεια των συγκεκριμένων αγορών. Η έννοια της αστάθειας έχει περιληφθεί και σε προηγούμενα σχέδια. Και είναι τελικά. Αυτό ακριβώς. Στο, RT, στο RTS 21 λέμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και το μέγεθος των συμμετεχόντων στην, στις αγορές. Εσείς λαμβάνετε υπόψη τον αριθμό, όχι όμως βέβαια το μέγεθος. Και για την εξαίρεση hedging περιλαμβάνει αυτή η περίεργη έννοια ότι βλέπουμε σε πολλά νομοθετήματα το hedging χαρτοφυλακίου, portfolio hedging. Όταν το χρησιμοποιείτε αυτή, αν χρησιμοποιήσω μάλλον την έκφραση αυτή, μπορεί κανείς να χωρέσει εκεί μέσα οτιδήποτε. Και δεν βλέπω για ποιο λόγο το portfolio hedging να εξαιρεθεί. Μπορώ να συνεχίσω βέβαια και με άλλα, αλλά νομίζω ότι θα κατανοήσατε ότι δεν μας αρέσουν αυτά που μας έχετε υποβάλει. Έχουμε βεβαίως σεβασμό για την ΕΣΜΑ και τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, αλλά εν προκειμένου δυστυχώς, δυστυχώς θεωρώ ότι δεν εξυπηρετείται τον νομοθέτη, μάλλον εξυπηρετείται τα συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και εν τέλει δεν σας πληρώνουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Φέρμπερ. Πρώτα η ΕΣΜΑ και μετά η Κομισιόν. Στίβεν. Ευχαριστώ. Ήδη το έχουμε πει ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Κυρίως το θέμα της καθυστέρησης, της αναβολής. Σίγουρα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε μαζί σας. Είτε σε scrutiny slot όπως τώρα, είτε σε κάποια άλλη μικρότερη συμμετοχή ή συνάντηση. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις μετά την υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών το Σεπτέμβριο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και γραπτά αυτή την εβδομάδα ακόμα. Πρώτα απ' όλα, γενική παρατήρηση, θέλω να σας πω ότι η MIFID 2 αποτελεί μια τεράστια αλλαγή. Υπάρχουν στοιχεία για τα οποία δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους επενδυτές, για τις κεφαλαϊκές αγορές θα έπρεπε να ξαναδούμε τις τεχνικές προδιαγραφές όταν θα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Δεν λέω ότι δεν δουλεύουμε ήδη σε αυτό το στάδιο για τις καλύτερες προδιαγραφές όσον αφορά το RTS, αλλά λέω ότι οι επιπτώσεις της MIFID 2 θα είναι τέτοιες που θα απαντηθούν αργότερα και θα πρέπει να δούμε πώς τελικά οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές, τα regulatory technical standards, θα λειτουργήσουν όταν έχουν τεθεί σε εφαρμογή και μετά θα επιστρέψουμε στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία έγκριση. Επιτρέψτε μου τώρα για την καθυστέρηση να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι τις επικρίσεις σας. Ε, φυσικά, ούτε κι εγώ είμαι ευτυχή που χρειάζεται να σα μιλήσω για καθυστέρηση. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Ούτε ρυθμιστέ θέλουν να καθυστερήσουν. Αντίθετα, θέλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να μπουν σε εφαρμογή κανόνε. Όμω είμαστε αντιμέτωποι με μια συγκεκριμένη πραγματικότητα για την οποία ήθελα να σας μιλήσω. Εννοείται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση πάντως θα είναι απόφαση των συνομοθετών. Δύο στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την καθυστέρηση αυτή. Πρώτον, οι λόγοι εξαρτώνται από την τελική μορφή των RTS. Ήδη το είπα και στην αρχή ότι εμείς πιστεύουμε πως η καθυστέρηση έχει να κάνει κύρια με τις αλλαγές, τη διαφάνεια και τα όρια θέσεων. Εκεί είναι που αργήσαμε να αποφασίσουμε όσον αφορά το περιεχόμενο. Εξαρτάται λοιπόν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές πώς θα προχωρήσουν, θα εξαρτηθεί και η καθυστέρηση. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από την ουσία, αλλά από πιο περίπλοκες ε, ρυθμίσεις των RTS. Γι' αυτό και θα υπάρχουν επιπτώσεις στην ε, εκπόνηση των ε, συστημάτων πληροφορικής. Τα είπα και στην αρχή. Και εδώ υπογραμμίζουμε, αλλά και σε κάθε συζήτησή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με θέματα συλλογής στοιχείων μέσω πληροφορικής. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους επόπτες, έχουν να κάνουν και με τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και με τις ε, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Προσπαθούμε βέβαια να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Ακούμε τις συζητήσεις που γίνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές, τα RTS, και ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνίες, το 2016 δηλαδή. Οπότε, δεδομένου ότι πρέπει να έχετε τα σωστά συστήματα, και επαναλαμβάνω δεν πρόκειται μόνο για τους ρυθμιστές, δεν πρόκειται μόνο για την ΕΣΜΑ, πρόκειται για τα πληροφορικά συστήματα των πλατφόρμων διαπραγμάτευσης με τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί καλά. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο για αποπτικούς λόγους, για να καταλάβουμε τι γίνεται στις χρηματοοικονομικές αγορές, αλλά τα στοιχεία αυτά τα χρειαζόμαστε ώστε η αγορά να μπορεί να λειτουργεί. Πρέπει τα συστήματα αυτά πληροφορικής να τα έχουμε ήδη για να καθορίσουμε ποιο ομόλογα έχουν ρευστότητα και ποια δεν έχουν. Άρα δεν πρόκειται μόνο για αποπτικού λόγους ή για να κατανοήσουμε καλύτερα την αγορά. Τα δεδομένα αυτά χρειάζονται για να μπορέσει η αγορά να λειτουργήσει. Συνεπώς, μαζί με αυτό τον παράγοντα, λειτουργίας αγοράς δηλαδή, ξέρουμε ότι τα συστήματα πληροφορικής αυτά μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούνται όταν θα ξέρουμε τις λεπτομέρειες για το RTS. Τότε μπορείτε να αρχίσετε να φτιάχνετε τα συστήματα πληροφορικής. Θέλω να υπογραμμίσω ότι λυπούμεθα που σας φέρνουμε αυτό το μήνυμα της καθυστέρησης, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πρακτική διαπίστωση, μια πραγματικότητα που μας κάνει να είναι πάρα πολύ δύσκολο 1η Ιανουαρίου να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται αναβολή. Τώρα και δύο άλλα θέματα ουσία θέλω να σχολιάσω παρακαλώ. Και ε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τα σχόλια που μας δώσατε. Λοιπόν, για το πώς ε, μετρούμε την ρευστότητα. και τα 100.000 ευρώ όρια για καθημερινές συναλλαγές και το 8%. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι συσσωρευτικό. Δύο μέρες δεν φτάνουν από μόνες τους. Πρόκειται για το συνδυασμό των δύο μερών με τις 100.000 και το 80% των ημερών και 100.000, αυτά τα δύο, που συσσωρευτικά πρέπει να υπάρχουν. Βάσει αυτού, μόνο 5% της αγοράς ομολόγων θα υποβάλλεται στις προδιαγραφές ε, διαφάνειας, στις απαιτήσεις διαφάνειας. Μπορείτε φυσικά να έχετε πιο στερεές απαιτήσει. για περισσότερες ημέρες, αλλά πάντα εξαρτάται από τον αριθμό των ομολόγων που θα υποβάλλονται στο καθεστώς διαφάνειας. Οπότε το καθεστώς αυτό χρησιμοποιώντας αυτά τα μέτρα θα καταλήξει στο 5% της συνολικής αγοράς ομολόγων που θα υποβάλλονται στις απαιτήσει διαφάνειας. Πρέπει να είμαστε και επιστοί στους στόχους του νομοθέτη. Περισσότερη διαφάνεια στην αγορά ομολόγων δηλαδή. Τέλος, για τα όρια θέσεων. Ο Ροντρίκο μπορεί βέβαια να προσθέσει και άλλες λεπτομέρειες αυτά που θα πω εγώ. Ακούσαμε διάφορες επικρίσεις. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο τεχνικό σημείο. Πράγματι, υπάρχουν διαφορές με την Αμερική. Πόσο διαφορετικό είναι το σύστημα. 28 συμβάσεις έχει η Αμερική. Εδώ πέρα μιλάμε για χιλιάδες ευρωπαϊκές συμβάσεις που πρέπει να υποβάλλονται στο σύστημα αυτό. Και επιπλέον, ο Αμερικανός ρυθμιστής μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα αναβδομάδα στις ε, θέσεις που επιβάλλει στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ενώ σε εμά θα χρειάζονται 9 μήνες αν περάσουμε μέσα από το σύστημα RTS. Και πρέπει να έχουμε και τη σωστή ισορροπία. Να διασφαλίζουμε δηλαδή ότι δεν γίνεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέση στην αγορά παραγόγων και από την άλλη μεριά να υπάρχει ρευστότητα σε μικρές αγορές και να διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας των ορίων θέσεων. Επίσης υπήρχε ένα σύστημα με πληροφορίες για χρόνια όσον αφορά τα όρια θέσεων, τις θέσεις πρώτα απ' όλα με διαφάνεια. Και μετά εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί στην Αμερική. Εδώ απευθείας βάζουμε τα όρια στην Ευρώπη. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτό το εύρος. Αν τώρα μέσα σε κάποιες περιόδους φανεί ότι έχουμε περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία της αγοράς αυτής και θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικές απαιτήσεις, μπορούμε να το κάνουμε. Υπογραμμίζω πάντως και τονίζω ότι πρόκειται για χιλιάδες συμβάσεις και όχι για 28. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πληροφορίες για την τρέχουσα θέση και γι' αυτό πρέπει απευθείας να έχουμε το Το 25% τώρα είναι ένα σημείο αναφοράς. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι με την ΕΣΠΑ λέμε ότι έτσι κι χρειάζονται ε, γνωμοδοτήσεις πριν εφαρμοστούν τα νούμερα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό που θέλουμε είναι να μην προδώσουμε το στόχο του νομοθέτη και μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το εύρος του 5 με 35%. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Ροντρίγκο τώρα. Θα απαντήσω κι εγώ σε κάποια σχόλια. Γιατί Ορισμένες ερωτήσεις ε, τις, τις λάβαμε γραπτός και θα σας απαντήσουμε και γραπτός με περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, όμως θα απαντήσω σε κάποια ζητήματα στα σχόλια του κ. Φέρμπερ για τους πρώτους μήνες του καθορισμού ρευστότητας των χρηματοδοτών πιστοτικών μέσων θα μπορούσε να υπάρξει ένας κίνδυνος λάθος ταξινόμησης. Πάντως ξέρουμε ότι μια πρώτη ταξινόμηση των ομολόγων ή των παραγόγων μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ταξινόμηση στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Κατά την γνώμη μας αυτό θα διαρκέσει ε, ένα τρίμηνο το πολύ 5,5 μήνες. Τώρα, οι πρωτογενείς αγορές εξαιρούνται, ναι, γιατί στο πρώτο επίπεδο ζητείτε να ταξινομηθούν με βάση την ε, ε, τέτοια την, ε, την ε, κατανομή στο πρώτο επίπεδο. Τώρα, γιατί αποφασίσαμε το ISIN σε, για, για, την αναφορά των ε, συναλλαγών. Αυτό το έχουμε κάνει διότι οι απαιτήσει σημαίνουν ότι δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή σε ολόκληρη την αγορά, αλλά θέλουμε να πούμε τι χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας δουλειά. Ένα ενιαίο σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σε όλες τις χώρες και από όλους τους ε, επόπτες. Έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσουμε μία, ένα σύνολο προδιαγραφών και αυτό το εξηγούμε στην τελική μας ε, έκθεση λόγω του κάλυψης, ότι δεν είναι κερδοσκοπικό, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια εμπορικά συμφέροντα σε αυτό το θέμα, υπάρχουν κάποιες ανταγωνιστικές ε, ανταγωνιστικά μάλλον συστήματα. Εμείς θέλουμε να είναι λειτουργικό καθημερινά ε, για το στόχο της ρύθμισης της αγοράς και πιστεύουμε ότι το icing είναι το καλύτερο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι δυνατόν ήδη να χρησιμοποιηθεί για πολλά για πολλά και πολλές συναλλαγές και εμπορία προϊόντων. Ούτως ή άλλως τα OTC δεν αφορούν την MIFID. Όπως ξέρετε υπάρχουν άλλα παραδείγματα χρήσης του icing ως προαπέτηση Πρόσφατα το δεχτήκατε στο SFDR ως απαιτόμενο δίκτυ, ε, μάλλον ε, απαιτούμενη ταυτοποίηση στο πρώτο επίπεδο. Τώρα όσον αφορά το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς, ο κ. Φέρμπερ θα μας ρώτησε αν θα έχουμε στοιχεία για το πόσο μεγάλη είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έχουμε, όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, τη δυνατότητα, αλλά θα το κάνουμε ωστόσο, ακόμα και αν δεν είναι επί τη βάση επισήμων στοιχείων, θα δημοσιεύσουμε στοιχεία που βοηθούν τους εταίρους να ε, εκτιμήσουν το μερίδιό τους στην ε, αμερικανική αγορά. Τώρα, κατά πόσο υπάρχει στόχος ή σκοπός να ε, ορίσουμε με βάση τη γαλλική υπόθεση, το γαλλικό καθεστώς. Το γαλλικό καθεστώς ε, υιοθετήθηκε 9 μήνες πριν να συμφωνήσετε στο πρώτο κείμενο με στόχο την μετάβαση σε ένα ομοιόμορφο σύστημα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το, γερμαν... το γαλλικό σύστημα δεν εξαιρεί το hedging, άρα δεν είναι συμβατό με το... αυτό το σύστημα που θέλετε εσείς. Άρα όλοι οι υπολογισμοί γίνονται επί διαφορετικής βάσης. Ε, το 38 είναι ένα σημείο εκκίνησης ενός ε, μιας καθοδικής πορείας, όταν δηλαδή πρόκειται να εκπνεύσει μια σύμβαση. Δεν συμπεριλαμβάνει το hedging, άρα πιστεύουμε ότι δεν είναι, δίκ, ε, ε, δεν είναι απόδειξη για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα στο μέλλον. Υπάρχει ένα σχόλιο όσον αφορά την οικονομική ρευστότητα και τον ορισμό αυτής και κατά πόσο είναι εξαιρετικά ευρύς. Ναι, μάλιστα, συντομεύω. Είναι δυνατό, ε, αδύνατο να έχουμε μια οικονομική, ε, τον ορισμό της οικονομικής ρευστότητας όπως ζητάτε. Αν είναι εξαιρετικά στενός μπορεί να παρακαμφθεί μέσω ενός εναλλακτικού ορισμού ή αν είναι πολύ ευρύς να μπορούμε πάλι να το παρακάμψουμε εντάσσοντας συμβάσεις μέσα σε αυτόν τον ορισμό. Ένα από τα δύο δεν μπορούμε να το τηρήσουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Εμείς ε, για λόγους σύνεσης έχουμε φτιάξει τον ορισμό πιο ε, περιοριστικό. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν θα καλύψουμε ποτέ τον τομέα που χρειάζεται να καλυφθεί. Τέλος, το θέμα του hedging των χαρτοφυλακίων το χαρτοφυλακείο hedging θα πρέπει αυτό να γίνει ε, με ακρίβεια σχετική και γι' αυτό και οι συναλλαγές που δεν είναι hedging δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Και γι' αυτό και τηρούμε το άρθρο 5 του RTS. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάω και το χρόνο. Ε, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος ακούσαμε με πολύ προσοχή τις ε, παρατηρήσεις και τις ανησυχίες σας. Ακούσαμε επίσης τις απαντήσεις της ΕΣΜΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα όρια θέσεων και τη διαφάνεια και τη ρευστότητα στην αγορά ομολόγων και όλα αυτά είναι εξαιρετικά ε, σημαντική συμβολή στην εσωτερική διαδικασία ελέγχου που έχει ξεκινήσει ε, Τώρα βέβαια θα πρέπει να αποφασίσετε για το τι έχει φτιάξει η ΕΣΜΑ με σεβασμό της απόψεις του Κοινοβουλίου. Εάν θέλουμε να καθυστερήσουμε την ΜΕΦΙΤ 2, ο στόχος είναι να αλλάξουμε μόνο την ημερομηνία. Κανείς δεν θέλει να αναλάβει τον κίνδυνο του να ακυρωθεί η συμφωνία την οποία πέτυχε οι νομοθέτες. Τώρα όσον αφορά τη διάρκεια της καθυστέρησης θα πρέπει να μην είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή. Γιατί αν ε, δεν καθυστερήσουμε επαρκώς, ε, κινδυνεύουμε για λόγους πληροφορικής ε, να καθυστερήσουμε μια δεύτερη φορά και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Άρα λοιπόν αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να το να αποφύγουμε. Από την άλλη πλευρά βέβαια αν καθυστερήσουμε υπερβολικά πολύ εξ αρχής ε, μπορεί να χάσουμε την κατάλληλη ευκαιρία και τελικά ο κόσμος να μην ασχοληθεί πλέον με τα αυτά που θα πρέπει να εκπονήσει. Είτε είναι οι εθνικές αρχές είτε είναι ο κλάδος που στοχεύουμε. Πρέπει να βρούμε δηλαδή μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της καθυστέρησης, η Κομισιόν θα το συζητήσει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την ΕΣΜΑ και θα ήταν καλή ιδέα να γίνει μια άτυπη συνεδρίαση σύντομα ώστε να μπορέσουμε πώς θα, να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, Φάμπιο, ή επειδή θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις, ναι η ερώτησή μου ε, δεν απαντήθηκε. Από πότε ξέρετε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση, ότι υπάρχει ανάγκη για καθυστέρηση και πότε ενημερώσατε την Κομισιόν. Κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησα να τονίσω σε σχέση με το μέγεθος του ζητήματος είναι ότι ε, θα ε, ξέρουμε καλύτερα όταν θα αποφασίσουμε τελικά για το RTS, για τις τεχνικές προδιαγραφές. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να ενημερώσουμε. Δύο εβδομάδες μετά από την ε, δική μας συνεδρίαση, άρα πριν από ένα μήνα έγινε αυτό μόλις. Ευχαριστούμε. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκα. Θα κοιτάξω να οργανώσω συνάντηση με την πραγματευτική ομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετείχατε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση και την ΕΣΜΑ και την Επιτροπή. Βέβαια, τα νέα που μας φέρατε δεν ήταν όλα πολύ καλά όσον αφορά το πλαίσιο, τη διαδικασία, αλλά για το περιεχόμενο, μια που έχετε πολλές ε, επιστολές και παρατηρήσεις από συναδέρφους, να τα λάβετε υπόψη σας και θα έχουμε και εκείνη η επιστολή από την πραγματευτική ομάδα. Και θέλουμε απαντήσεις γραπτά στις ερωτήσεις μας. Είναι πάντα προτιμότερο από το να μας δίνετε μόνο προφορικά τις απαντήσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμός και σύγκληση στις πολιτικές στον τομέα της φορολογίας των εταιριών στην Ένωση. Δύο εισηγητές έχουμε εδώ, την Αναλίζε Ντότς και Λούντεκ Νίτερμαγερ. Ποιος θα αρχίσει? Αλλιώς θα αποφασίσω εγώ. για μένα είναι η έκθεση Dodge Niedermayer, συνεπώς αναλύζει. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ελπίζω την επόμενη φορά να αρχίσει ο κύριος Niedermayer για να υπάρχει ισοτιμία μεταξύ μας απόλυτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Niedermayer και το προσωπικό και τη γραμματεία και όλους τους σκιώδεις εισηγητές Ευχαριστώ επίσης και όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες στο κείμενο. Εννοείται ότι υπήρχαν πάρα πολλές τροπολογίες και ευχαριστώ πολύ όλους σας. Η διαδικασία πάντως αυτή τροπολογιών έκανε, κατέδειξε το ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές απόψεις στο Κοινοβούλιο και για να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό προσπαθεί να κάνει, γι' αυτό και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για τη διαδικασία και ο κύριος Νίγη Ντεμάγερ σίγουρα θα συμπληρώσει. Η Γραμματεία έχει δουλέψει σκληρά για να καταλήξει σε συμβιβαστικές τροπολογίες, είτε μέσω του κειμένου, και καταλαβαίνετε ότι πάντα όταν υπάρχουν τόσο πολυάριθμες τροπολογίες, πολλές φορές επαναλαμβάνονται και γι' αυτό πρέπει να γίνονται και αλλαγές για να κρατάμε τη συνοχή του κειμένου. Να είσαστε λοιπόν παρακαλώ υπομονετικοί, να δείξετε κατανόηση τώρα που προσπαθούμε να συμμαζέψουμε κάπως τις τροπολογίες και να καλύψουμε όλους σας. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τομείς για τους οποίους έχουν υποβάλει τροπολογίες οι συνάδελφοι με σκοπό να ενισχυθεί το κείμενο. Πράγματι, φροντίζω κι εγώ με τη γραμματεία να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε δουλέψει πάνω στα παραρτήματα που καλύπτουν όλες τις συστάσεις που έχουν να κάνουν ε, με τις διάφορες κατηγορίες εκθέσεων. Μετά θα δούμε τις αιτιολογικές σκέψεις και τις συστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις τωρινές κατηγορίες. Σίγουρα χρειάζεται διευκρίνηση του κειμένου, όπως αφήνει Και πολλές τροπολογίες πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρίω για το θέμα αυτό του πεθετικού φορολογικού σχεδιασμού, για το θέμα των φορολογικών ρυθμίσεων, tax rulings. Υπάρχουν τομεί όπου χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές από τους συναδέρφους. Κάποιες τροπολογίες είναι για τους ελεύθερους λιμένες και θέλουμε να καταλάβουμε τι προσπαθούν να πετύχουν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου προσπαθούμε να πετύχουμε συμβιβασμό μεταξύ διαφορετικών θέσεων. Πολλών διαφορετικών θέσεων μερικές φορές που υποβάλλουν οι συνάδελφοι για θέματα όπως είναι το CCTB. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω και το συνεισηγητή μου και όλους τους σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους έχω μιλήσει ξανά και ξανά για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατόν συμβιβαστικές τροπολογίες που να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερες πολιτικές ομάδες. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια έκθεση η οποία έχει βάση. Οι ομάδες δηλαδή στο μεγαλύτερο βαθμό στηρίζουν την έκθεση αυτή και θα φανεί αυτό και στην ψηφοφορία. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον συνεισηγητή μου. Ευχαριστούμε Αναλίζε. Τώρα όντω, ο Λούντεκ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θέλω και εγώ να επαναλάβω ότι εκτιμάω απολύτως την προσπάθεια που έχει γίνει με τροπολογίε και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ την Αναλύσα για την συνεργασία της αλλά και την γραμματεία. Πολλέ τροπολογίε πράγματι μπορούν να βοηθήσουν να γίνει ακόμα καλύτερη η έκθεση γιατί διευκρινίζουν κάποια σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση και φροντίζουν να είναι πιο εύκολα κατανοητά. Υπάρχουν και τροπολογίες που θα είναι πιο δύσκολο να πετύχουν ευρεία υποστήριξη. Βέβαια, στη ψηφοφορία θα φανεί αυτό. Έτσι δουλεύουμε. Πάντως, για τις διευκρινήσεις έχουμε πολλές νέες ιδέες που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση των απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις εξετάζουμε Και ακόμα και σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να δούμε πώς θα τις συμπεριλάβουμε, εφόσον βέβαια πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση που πηγαίνει και η έκθεση γενικότερα. Όσον αφορά τη διαδικασία, όπως είπε και η Αναλύζη, ε, προσπαθούμε να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Το παράρτημα είναι το τμήμα αυτό της έκθεσης που είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί είναι που χρειάζεται νομοθετική δράση. Εκεί επικεντρωθήκαμε την ε, πρώτη φορά και την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε με τους σκιώδεις και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καταλήξει την επόμενη εβδομάδα σε μια πρώτη απόπειρα συμβιβαστικών τροπολογιών. Η συζήτηση με τους σκιώδες είναι πολύ σημαντική γιατί θέλουμε να έχουμε τη στήριξή τους. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για να έχουμε μια καλή έκθεση και έκθεση με συνοχή. Πάνω από 300 τροπολογίες υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν μείνουμε με τόσες πολλέ δεν θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο. Γι' αυτό και προσπαθούμε να πετύχουμε συμβαστικέ λύσεις. Η συνοχή και η ευκρίνεια του κειμένου θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στο προήμιο όσο ε, το παράρτημα. Έτσι έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την θέση μας, το Συμβούλιο και Επιτροπή και να, να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τη διάβρωση φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, το BEPS. Θέλουμε λοιπόν βελτίωση όσον αφορά τον φόρο των εταιριών και επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις ώστε το αποτέλεσμα να είναι σαφές και κατανοητό. Με συμβασμούς, δεν εννοώ συμβασμούς ανάμεσα στην αναλύση και εμένα ή τις ομάδες μας, αλλά συμβασμούς ώστε να έχουμε την ευρύτερη δυνατόν στήριξη. Συγχρόνως πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε ασάφειες μέσα στο κείμενο. Δηλαδή τροπολογίες που δεν είναι σαφείς ή που πηγαίνουν ε, πολύ πιο πέρα από το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τότε υπονομεύεται η σαφήνεια του κειμένου και ε, άρα και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει όσον αφορά ε, τα BEPS, τη διάβαση φορολογικής βάσης και μεταφορά κερδών. Προσπαθούμε λοιπόν, όπως σας είπα, για την επόμενη εβδομάδα να ετοιμάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες για να ψηφιστούν στην ΕΚΟΝ. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή έκθεση, μια καλή πρόταση με ευρεία στήριξη και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια. Προσβλέπω να συνεχίσουμε την επαφή με τους σκιώδες αλλά και όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές ώστε να συμπεριλάβουμε όσο γίνεται περισσότερο τις ιδέες σας στο κείμενό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στους ε, σκιώδεις από τις διάφορες ομάδες και τώρα ξεκινάμε με τον κύριο Λούτκε, ECR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ καταρχήν τους δύο εισηγητές για την εξαιρετική τους δουλειά. Είμαι ευτυχής που μπορώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους σε αυτή την έκθεση. Έχω θετική στάση απέναντι σε αυτή την έκθεση. Έχω όμως κάποιες τροπολογίες και θα σας τις εξηγήσω σύντομα. Καταρχήν, όσον αφορά τη σύσταση για το σήμα του έντιμου φορολογούμενου. Ε, ε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι ε, δεν είναι συμβατό με το απόρριτο της ε, φορολόγησης των εταιριών θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, δραστηριότητες lobbying απέναντι στις φορολογικές αρχές λόγω όλων αυτών. Δηλαδή ένας ε, αγώνας θα πρέπει να γίνει για να μπορέσει κανείς να έχει αυτή την αναγνώριση ως έντιμος φορολογούμενος. Και για να αποφύγει δηλαδή τους ελέγχους. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Έπειτα. Έχουμε την κοινοποίηση των προληπτικών φορολογικών συμφωνιών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να προβλέπετε να στέλνετε και στην Κομισιόν και στη Γενική Διαθέση για τον Ανταγωνισμό, γιατί δεν πρόκειται μόνο για φορολογικά θέματα, αλλά και για την πρόληψη ενδεχόμενων παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό η Κομισιόν να έχει σχετικές, τις σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Θα πρέπει λοιπόν και η Κομισιόν να είναι ανάμεσα στους παραλήπτες αυτών των πληροφοριών. Η αξιολόγηση τώρα των της απώλειας ε, και ε, κερδών νομίζω πως είναι προβληματικό μέσο. Ε, Διότι διαβλέπω τον κίνδυνο πολιτικοποίησης και ούτως ή άλλως αυτή η φόροι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα βρίσκω ότι υπάρχει και κενό νομιμοποίηση Από τη δική μας λοιπόν πλευρά, εμείς ζητούμε διαγραφή. Όσον αφορά τώρα την κοινή φορολογική βάση εταιρική φορολόγηση, η ομάδα μας, η CR, επίσης ζητεί διαγραφή της προτάσεως, θεωρώντας ότι είναι θέμα φορολογικής κυριαρχίας των χωρών μελών. Σα τα εξηγώ αυτά ως εκπρόσωπο τη πολιτική μα ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών ε, και Μεταρρυθμιστών. Προσωπικά ωστόσο σημειώνω, θεωρώ εγώ ότι η ενιαία φορολογική βάση για την φορολογική εταιριών είναι σωστή βάση και ιδίως τα στοιχεία μιας ενοποιημένης φορολογικής βάσεως και μιας υποχρεωτική, ε, υποχρεωτικού μάλλον τρόπου υπολογισμού είναι σημαντικά και δεν αποδυναμώνουν τα εθνικά μέτρα. Εφόσον δεν πρόκειται για ε, ε, ρύθμιση εκ μέρους της Ευρώπης των, ε, ε, του τρόπου υπολογισμού του φορολογικού συντελεστού. Γι' αυτό ε, θα κάνω εγώ μια προσωπική τροπολογία που να λέει ότι πρέπει να αποφευθεί αυτό εφόσον μικρές και μεσές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν και η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να αναφέρεται στον ορισμό της βάσης και αυτό είναι επαρκές. Και θα πρέπει να υπάρχει, να ισχύει μάλλον το ίδιο δίκαιο για, την, για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης για όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα για την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που προτείνεται να αποσπαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να γίνει ανεξάρτητη αρχή για να εξασφαλίζεται και η ανεξαρτησία της, ε, των σχετικών ελέγχων. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η τροπολογία που απευθύνεται στην σύσταση Β2. Εμείς προτείνουμε επίσης διαγραφή της πρότασης σε 1 για την σύναψη διεθνών φορολογικών συμβάσεων, διότι οι φορολογίες αυτές δεν είναι αρμόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας. Κάτι που θα μπορούσε να κάνει κανείς θα ήταν να λάβει μέτρα, ε, να εξετάσει μέτρα δικαστικής ε, δράσης για περίπτωση χρήσης φορολογικών παραδείσων. Εδώ προτείνουμε και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εάν εμπορικές συμφωνίες με χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως φορολογική παράδειση, αν τέτοιου λοιπόν είδους ε, διεθνείς συμβάσεις μπορούν να καταγγελθούν και να πάψουν να Άλλα μέτρα για το κλείσιμο των δημοσιονομικών των φορολογικών κενών δεν θεωρούμε να είναι ορθά, διότι πάλι εδώ θέμα συγκρούσεως αρμοδιοτήτων. Διότι οι αρμοδιότητες αυτές είναι αρμοδιότητες του εθνικού επίπεδου και θα πρέπει αυτά να εξαιρεθούν από το κείμενο, διαγραφούν από το κείμενο της εκθέσεως. Τέλος, θα πρέπει να καταληφθούν τα θύματα εκείνα της εκθέσεως που δεν αναφέρονται στον ε, φόρο, στη φορολόγηση δηλαδή εταιριών, αλλά έχουν σχέση με τον ΦΠΑ, διότι αυτά εκφεύγουν από το πεδίο της εκθέσεως αυτή θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην φορολόγηση επιχειρήσεων και να μην υπησέλθουν άλλα θέματα άλλων φόρων. Και βεβαίω πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα όρια αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν αυτά. Σα ευχαριστώ κύριε Λούκε. Φιλελεύθερη ε, ομάδα, ομάδα φιλελευθέρων μάλλον. Δεν βλέπω να είναι παρούσα εισηγήτρια. Ούτε και βλέπω άλλους. Μακάρθη από την Ενωτική Αριστερά. Α, επίσης απόνοια, πούσα. Α, εδώ είστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες και όλοι θα αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουση. Ορισμένοι από εμά έχουμε πιο συγκεκριμένε ιδέε για ορισμένα από τα στοιχεία της συγκρούσεως αυτή. Δύο κέρια θέματα για τον φόρο εταιριών. Να πληρώνουν δίκαιο τμήμα που να ανταποκρίνεται, δηλαδή που να ε, είναι σύμφωνο με τα έσοδά τους η επιχείρηση. Και βεβαίως το άλλο θέμα είναι το ζήτημα της επικουρικότητας ή της κυριαρχίας των χωρών μελών. Στις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει κάνουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση και την διόρθωση της ισορροπίας αυτής. Πρώτα δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουν ενδιαφέρον για τους πολίτες αλλά και για τις να καθίστανται δημόσιο κτήμα με τον εντονότερο δυνατό τρόπο να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες και αφετέρου να προστατεύονται τα δικαιώματα των κυβερνήσεων να θέτουν τα δικά τους φορολογικά όρια και για τον εταιρικό φόρο, την εταιρική φορολογήση δηλαδή. Βλέπουμε ορισμένε κυβερνήσεις και την Ιρλανδική κυβέρνηση να επαναφέρουν συστήματα τα οποία θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποφεύγουν την καταβολή του αναλογούντος φόρου. με τα σχετικά νομοθετήματα που καταθέτει δηλαδή στην ε, Ιρλανδική Βουλή ή η Ιρλανδική Κυβέρνηση. Οι μηχανισμοί στους οποίους θα προσφεύγουν οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι γνωστοί στους πολίτες και να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσοι φόροι εισπράττονται και ε, πόσα από τα έσοδα αυτά καταλήγουν σε δημόσιες υπηρεσίες. να γίνονται δε σεβαστά τα, τα κυριαρχά δικαιώματα των κυβερνήσεων. Και εφόσον θέλουν να αυξήσουν τον φόρο των εταιριών, να το αυξήσουν. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμά, γραμμή, συγγνώμη, απολύτως για μας. θα επιζητήσουμε και συμβαστικές τροπολογίες ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο εκθέσεως που να μπορούμε να το υποστηρίξουμε συλλογικά έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει κείμενο το οποίο να το υποστηρίζουν και οι ψηφοφόροι μας. Προσοχή λοιπόν. Υπάρχει το ενδεχόμενο οι μεγάλες πολιτικές ομάδες να συνεργαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την προσπάθεια αυτή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι λάθος, διότι τότε ό,τι και να ψηφίσει το Κοινοβούλιο, θα το απορρίψουν οι κυβερνήσει στο Συμβούλιο και ίσω και δικαίω. Και ίσω να το απορρίψουν και οι πολίτε οι ίδιοι. Μάλιστα, σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Μόλι των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ και τους δύο εισηγητές για την σκληρή του δουλειά και για την καλή σχέση που έχουμε σε έναν δύσκολο τομέα όπου υπάρχουν διαφωνίες και μέσα στην ίδια ομάδα αλλά και μεταξύ ομάδων. Οπότε είναι ένα δύσκολο θέμα, δύσκολο θα επιληθεί. Αρχίζω με κάποια σχόλια επί της διαδικασίας πριν μπω στο περιεχόμενο των τροπολογιών μας. Αρχίσαμε με διάφορες συναντήσεις διμερείς και σκιωδών, κάτι που ήταν πολύ επικοδομητικό πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά από τη στιγμή που πήραμε την έκθεση δεν έχουμε συναντήσεις σκιωδών. Τις επόμενες εβδομάδες βέβαια θα υπάρξουν. Η Αναλίζα είπε ότι τους συμβασμούς τους κάνει η γραμματεία. Εγώ όμως, αλλά και άλλες ομάδες, ανησυχούμε, γιατί φοβούμαστε ότι θα καταλήξουμε σε σεβασμούς μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων. Και αν γίνει αυτό, αυτό αντιβαίνει στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι όλες οι πολιτικές ομάδες να συμμετέχουν στην ε, διατύπωση συμβιβασμών και όχι μόνο οι μεγάλες. Αυτό λοιπόν θέλω να το υπογραμμίσω. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες, όπως είπε και η Αναλίζα και υπάρχουν διαφορές και μέσα στις ίδιες τις πολιτικές ομάδες, μέσα στην ίδια πολιτική ομάδα, πιο σωστά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν γραμμές αναχώρα μέλη, που ακολουθούν δηλαδή κάποιες χώρες και άλλη γραμμή κάποιες άλλες χώρες, που δεν είναι αυτό το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να καταπολεμήσουμε, ώστε να λειτουργούμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους και όχι των πολιτών της μιας ή της άλλης χώρας. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε το... Δεν θέλουμε το διέρη και βασίλευε. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η διαίρεση βάση εθνικών προτεραιοτήτων και αυτό να είναι πάνω από τα συμφέροντα της Ευρώπης ολόκληρης. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι πιστεύουμε πως ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται μεταξύ επιχειρήσεων βάσει καινοτομίας προϊόντων και υπηρεσιών και να μην ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις ή οι χώρες μέλη μεταξύ τους βάσει φορολογικών ρυθμίσεων. Δεν είναι αυτό που πρέπει να έχουμε σε μια Τώρα, επί της ουσίας για τις τροπολογίες μας, κάτι που δεν καλύπτεται καθόλου στην έκθεση είναι το θέμα των μεγάλων επιχειρήσεων και νομικών επιχειρήσεων. Η φοροαποφυγή είναι κάτι από το οποίο υποφελούνται τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ πρέπει να έχουμε τροπολογίες ισχυρές ώστε να σταματήσει η πρακτική αυτή των λογιστικών εταιριών. Έχουμε 314 για παράδειγμα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα και ε, στα συμφέροντα. Η δουλειά μας πάντως δεν είναι να συζητάμε με την Επιτροπή για αδύναμες προτάσεις, αλλά να τα βάζουμε τις χώρες μέλη που εφαρμόζουν κάποια μέτρα που πιστεύουμε εμείς ότι δεν είναι σωστά. Χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία με την πρόταση αυτή και να πιέσουμε περισσότερο την Επιτροπή όσον αφορά την κοινή ενωπημένη βάση φορολογία εταιριών, το CCTB. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοιες τροπολογίες, να δείξουμε ότι εμείς ηγούμεθα και όχι ότι ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, εμείς έχουμε ηγετικό ρόλο εδώ και εμείς με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στο Συμβούλιο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους καταγγέλλοντες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Επιτροπή για τις Φορολογικές Ρυθμίσεις δεν θα είχε υπάρξει αν ήμασταν σε πιο αδύναμη θέση και δεν είχαμε τις πληροφορίες που είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες και αυτό να αναφέρεται στην έκθεση. Ήδη υπάρχει κάποια προστασία, αλλά θέλουμε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στην τελική έκθεση. Τέλος, για τις εκθέσεις αναχώρα. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι θετικό, χαιρόμαστε που υπάρχει. Είναι κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε. Έτσι συνεισφέρει το Κοινοβούλιο στη διαφάνεια όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Τώρα, όπως είπα και πριν, χαίρομαι που θα έχουμε τρεις συναντήσεις μεταξύ σχεδόν εισηγητών και θα ήθελα να επιστρέψουμε στο πνεύμα των συμβιβασμών μεταξύ όλων και όχι μεταξύ των ε, μεγάλων πολιτικών ομάδων. Άλλο είναι οι συμβασμοί, άλλο είναι η συνένεση πλήρης ε, συνένεση είναι δύσκολο να επιτευχθεί και δεν είναι αυτό που προτιμάω, γιατί έτσι δεν θα προχωρήσουμε αρκετά. Ο πρόεδρος Φέρμπερ, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάτω. Μάρκο Ζάνη της EFTD. Σας ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ τους δύο εισηγητές που ξεκίνησαν έναν επικοδομητικό διάλογο. Ήδη έχουμε συγκεντρωθεί όλοι μαζί μια φορά και προέκυψαν σημαντικά στοιχεία προς συζήτηση, αλλά και κάποια σημαντικά στοιχεία επί των οποίων θα μπορούσε να βρεθεί κοινή συμφωνία. Άρα λοιπόν η κίνηση είναι εξαιρετικά θετική όσο με αφορά. Εγώ σύντομα θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα σημεία που κατά με είναι σημαντικά και που θα ήθελα να τονιστούν και στις ε, ε, συμβιβαστικές που θα συζητηθούν Καταρχήν πιστεύω ότι τα δύο πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να τονιστούν είναι η έννοια της διαφάνειας και αυτό σήμερα αποτελεί το θεμέλιο όταν μιλάμε για αυτό το πρόβλημα και κυρίως όσοι συμμετέχουν στις εργασίες ε, της Επιτροπής ΤΑΚΣ θα γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να ε, δούμε κείμενα και να πάρουμε πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Θεωρώ λοιπόν πως μια ένοπιτική προσέγγιση θα πρέπει να είναι αυτή της διαφάνειας. Ε, ε, μία αναχώρα ε, αναφορά που θα είναι δημόσια και που θα προσπαθήσει έτσι να θεσπίσει ένα πλαίσιο απλής ανάγνωσης ε, γιατί συχνά κυρίως το θέμα της ρύθμισης για την αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων στο ιστορικό μεγάλων επιχειρήσεων ή τραπεζών ή ομίλων αυτό το είδος η αποκάλυψη στοιχείων γίνεται με πολύ περίπλοκο τρόπο ενώ η δημοσίευση απαγόρευση των αναχώρα αναφορών είναι πολύ σημαντική, αλλά το εξίσου σημαντικό είναι το να έχουμε ένα πλαίσιο απλό, ευανάγνωστο, όχι μόνο για τους τεχνικούς δηλαδή, αλλά και για τον απλό πολίτη. Έπειτα πρέπει να δημιουργηθούν κοινέ προποθέσει ανταγωνιστικότητα για όλα τα είδη επιχειρήσεων στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν πω μια ισχυρή προσέγγιση που θα ενισχύει την αδύναμη προσέγγιση της επιτροπή για την ε, CCCTB είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προδιαγραφέ, κοινέ για όλε τι χώρε τη Ένωση και μετά να αφήσουμε κάποια διακριτικότητα στις ε, επιμέρους κυβερνήσεις για να ε, φτιάξουν ε, την φορολογία τους για τις επιχειρήσεις αλλά η φορολογική βάση θα πρέπει να είναι κοινή έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται οποιαδήποτε χώρα οποιαδήποτε εταιρεία αποφασίσει να εγκατασταθεί στην τάδε ή την χώρα. Τώρα, εδώ η φορολογική βάση δεν είναι θέμα ε, ούτε είναι θέμα η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη, όπου δεν υπάρχει συντονισμός πάντοτε όσον αφορά στην διαφάνεια, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν σκόπιμο να ε, σωματεωθεί ένα αίτημα για την θέσπιση ενός δημόσιου ευρωπαϊκού αρχείου για πληροφορίες για τέτοιου τύπου. Δεν υπάρχει κάποιο συντονισμό μια κοινή βάση ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικές βάσεις δεδομένων συχνά δεν το αναφέρουν. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες. Μια ε, ένα λοιπόν ε, δημόσιο και διαφανές αρχείο θα ήταν σημαντικό. Κάτι ακόμα που λείπει το, κατά τη γνώμη μου εδώ είναι τα εξή δύο. Καταρχήν, ρόλος των τραπεζών. Προφανώς οι τράπεζες είχαν και έχουν ε, πολύ σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό μάλλον όσον αφορά την στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας και στην βοήθεια προς τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις να ε, αποφεύγουν την φορολόγηση μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες όπου η φορολόγηση είναι χαμηλότερη. Σε αυτή την έκθεση και στην έκθεση της ε, Επιτροπής ΤΑΞ έχουμε, κάνουμε πολύ λόγο για τον σύμβουλο φορολόγησης αλλά δεν μιλάμε για το ρόλο των τραπεζών. Πάντω, είτε είναι νόμιμες, είτε είναι παράνομες οι δραστηριότητε, περνάνε μέσω από τραπεζικέ συναλλαγές. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε οι τράπεζε που λειτουργούν εντό τη Ένωση να λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί ε, αν μπορούσαμε να βρούμε τη ροή των χρημάτων, την πορεία των χρημάτων, κανένα δεν θα μπορούσε να κρύψει από πού προέρχονται, ούτε να φοροδιαφύγει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην κρύβουμε πια το ρόλο που παίζουν οι τράπεζες σε αυτή την υπόθεση. Κάτι ακόμα, αλλά από αυτού νομίζω θα είναι δύσκολο να βρούμε κάποια συμφωνία, αλλά θα ήθελα να το τονίσω, είναι ότι καθημερινά προκύπτει ότι υπάρχει ε, μέχρι και σήμερα σαφής πολιτική βούληση ορισμένων εκπροσώπων και ορισμένων κρατών μελών να μην θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα αυτό. Το νέο που ανεφέρθη πριν από λίγες μέρες για, σε κάποιες εφημερίδες της, Γερμανία, της Γερμανίας είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη μπλοκάρισαν στο Συμβούλιο ε, αποτελεσματικά μέτρα όσον αφορά τα tax ruling, τις ειδικέ ε, αυτές ευνοϊκές ρυθμίσεις, φορολογικές ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε Ποιο ακόμα και σήμερα δεν θέλει να λύσει αυτό το πρόβλημα και θέλει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, ε, έναν τρόπο που σαφώς δεν μπορεί πλέον να συνεχίζεται. Τελευταία παρατήρηση είναι ότι ε, προφανώς χρειάζονται συστάσεις όσον αφορά τον έλεγχο αλλά και τις κυρώσεις για όσους δεν σέβονται αυτούς τους κανονισμούς. Ε, συγκεκριμένοι ορισμοί δηλαδή, συγκεκριμένοι ορισμοί για τους φορολογικούς παραδείσους, για τη μαύρη λίστα και ένα φάσμα κυρώσεων δηλαδή με σταδιακό τρόπο για τις επιχειρήσεις και τους ομίλους που δεν σέβονται τους κανόνες διαφάνειας και που δεν συνεργάζονται και ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν σε χώρες ε, ε, της Ένωσης και που μπορεί να μπουν δηλαδή στους καταλόγους, ε, στις μαύρες λίστες. Τώρα, για τους πληροφοριοδότες, το έχουμε πει ότι και χωρίς τη δική τους παρέμβαση σήμερα εμείς δεν θα ήμασταν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε η ολόκληρη Ευρώπη θα μιλούσε για αυτά τα θέματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει μια πρόταση έτσι ώστε η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να θεσπίσουν ένα, μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα προστατεύει σοβαρά αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ ως Ιταλός ε, ε, θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση γιατί έχουμε νομοθεσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως best practice, καλύτερη πρακτική. Έχουμε εξαιρετική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία μαρτύρων ε, ε, που έχουν καταθέσει κατά της μαφίας. Μια τέτοια νομοθεσία λοιπόν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ΕΝΕΦ δεν βλέπω κανένα, από την ομάδα δηλαδή ε ΕΝΕΦ. Άλλος κανείς δεν ζητεί το λόγο. βλέπω, ναι, ναι, κάποιον. Κύριε Φερνάντες, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές, τον Λούντε και την αναλύση. Και θέλω να μιλήσω εκ μέρους του αυτού μου για τον Ραμόν Χάμνερ, επειδή υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες. Κάτι που λείπει, πιστεύουμε, στις διάφορες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους φορολογικούς παραειδήσους, είναι ότι θέλουμε αντικειμενικά κριτήρια για να ορίσουμε ποιοι είναι αυτοί. Ο Ραμόν λοιπόν και εγώ έχουμε υποβάλει μια τροπολογία για να συμπεριλάβουμε κριτήρια που μπορούν βέβαια να αυξηθούν να μειωθούν. Προτείνουμε αν μη τι άλλο κάποια κριτήρια που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καθορίσουμε τι είναι φορολογικός παράδεισος. Κάνουμε προτάσεις λοιπόν. Χαμηλή φορολογία, η ανύπαρκτη, ε, προσφέρουν φορολογικές διευκολύνσεις σε ξένους, ε, που δεν έχουν οικονομικές δραστηριότητες εκεί, δεν δίνουν πληροφορίες, έχουν μυστικές συμφωνίες, δεν υπάρχει διοικητική συνεργασία ή αστυνομίας, ε, τραπεζικό απόρριτο, ε, προστασία σε κατακέλλοντες. Εν πάση περιπτώσει, για κάποια από αυτά τα σημεία είναι ένας κατάλογος που μπορεί να συμπεριλάβει και παραπάνω κριτήρια. Αλλά λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κατάλογο κριτηρίων για να ξέρουμε πότε έχουμε να κάνουμε με φορολογικό παράδεισο και πότε όχι. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Πώς θα εφαρμοστεί όμως. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια υπηρεσία που να αναλάβει να εντοπίζει και να καταγράφει τις περιπτώσεις tax ruling διασυνορικές ή όχι, να, υπάρχει, να έχει τον κατάλογο αυτό των φορολογικών παραδείσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια κλπ. Πιστεύω δηλαδή ότι η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας και να κοροϊδευόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνομοθετεί σε φορολογικά ζητήματα με το Συμβούλιο επίσης. Το Συμβούλιο Σόμπλε έχει πει εδώ στην Επιτροπή μας πριν από λίγο καιρό ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε κατά πόσο οι αποφάσεις πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται ομόφωνα ή όχι. Πας περιπτώσει αυτές είναι οι τροπολογίες μας και ευχαριστώ πολύ και την Αναλύζη και τον Λούντικ για το έργο τους. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Φέρμπερ. Α, εσείς κύριε Σάντ. Ορίστε. Ένα σύντομο θέμα. Προτείνω επειδή μία μικρή μειοψηφία ευρωβουλευτών έχουν κάπως ανάμεικτα συναισθήματα για το θέμα αυτό. Είμαστε μεν υπέρ της διαφάνειας, αλλά μας απασχολεί η σύγκληση. Στο τέλος του το κείμενο κάνει μια διάκριση ενιών μεταξύ των όσων περιλαμβάνει για διαφάνεια και όσα περιλαμβάνει για σύγκληση. Δηλαδή μπορεί να ψηφίζουμε υπέρ της διαφάνειας αλλά όχι απαραίτητα υπέρ της σύγκλησης. Ο συντονισμός είναι κάτι το μεικτό, δηλαδή συντονισμός για τη διαφάνεια, συντονισμός ε, φορολογικών πολιτικών. Αν πρόκειται για συντονισμό για τη διαφάνεια, καλώ. Αν όμω πρόκειται για συντονισμό ή σύγκριση, δηλαδή ε, να πάνε όλοι οι φορολογικοί συντελεστέ προ την ίδια κατεύθυνση, αυτό δεν μα βρίσκει σύμφωνο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια διάκριση μέσα στο κείμενο, έτσι ώστε και η ψηφοφορία να είναι ξεκάθαρη και διαφανή. Ευχαριστώ αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Φέρμπερ. Τότε θα δώσω το λόγο πάλι στου ε, εισηγητέ. Εσεί πρώτα κύριε Νίτερ Μάιερ. Πρώτα εξετίμησα ιδιαίτερα τη συζήτηση που έφυξε θέματα που θα μας απασχολήσουν και στις προσεχείς ημέρες. Η ε, συνάντηση των ε, σκιωδών θα πρέπει να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Αλλά ας αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Να προτείνουμε δηλαδή συμβαστικά κείμενα. Συμβασμό σημαίνει ότι ε, γίνεται αποδεκτή η διατύπωση από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Μόνο μέσω των συμβαστικών διατυπώσεων μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνεκτική έκθεση και όχι ψηφίζοντας 300 διαφορετικές τροπολογίες τη μια μετά την άλλη. Ελπίζω ότι θα συζητήσουμε όλα τα θέματα εδώ, επίσης τα ζητήματα της ουσίας και έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια και στο παράρτημα Τα προβλήματα των BEPS δεν έχουν προκληθεί από τον ΟΣΑ και τα G20. Και εμείς ζητήσαμε να, ζητήσαμε να συζητηθούν τα θέματα αυτά και πάνω από δύο χρόνια. Και αυτό που συζητούμε τώρα είναι πώς να βρούμε την καλύτερη απάντηση στα BEPS. Το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί εδώ και ε, καιρό. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον την συζήτηση, να μείνει ξεκάθαρη και ευνόητη η ε, διατύπωση της εκθέσεως και αυτό κυρίως μας ενδιαφέρει. Η κυρία Ντότζ, σας ευχαριστώ. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω η ενδήποτε συζήτηση θα διεξαγάγουμε στη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Αλλά χρειάζεται κάποια διευκρίνηση για ορισμένα θέματα. Πολλοί μας βοήθησαν τα σχόλια των συναδέλφων και σας ευχαριστώ. Σύντομα τώρα ο κύριος Λούκε έφυξε ορισμένα σημαντικά θέματα. Πρώτα, όσον αφορά την ετικέτα του έντιμου φόρου, του δίκαιου φόρου δηλαδή, πρέπει να το δούμε. Να δούμε τα κείμενα και πώς μπορούμε να κάνουμε το κείμενο πιο αποδεκτό. Όσον αφορά στο α6 και η προσπάθεια της Κομισιόν να υπολογίσει το ε, δημοσιονομικό κενό. Ήδη έχει πολιτικοποιηθεί το θέμα, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει μια πιο στέρεα διαδικασία, μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο από το πολιτικοποιημένο αυτό ε, χαρακτήρα, κάποιο, κάποιο στοιχείο από το πολιτικοποιημένο αυτό χαρακτήρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε κι άλλο όμως αν θέλετε. Το ζήτημα του ρόλου της Κομισιόν στις διεθνείς συμφωνίες, αναφέρομαι στο ΣΕ1, και λέω μόνο ότι αυτές οι εμπορικές ε, συμφωνίες καλύπτονται στο σε 3. Άρα λοιπόν το ζήτημα που λέτε ίσως να είναι ήδη μέσα στο κείμενο. Πρέπει να το συζητήσουμε. Τέλος για τις φορολογικές αμνηστίες. Φαίνεται να διαμορφώνεται κάποια επιθυμία από χώρες μέλη και άλλους φορείς ε, να λάβουν περισσότερες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να δίνεται αμνηστία χωρίς βέβαια να θέλουμε να μπούμε σε ε, ζητήματα κυριαρχίας των χωρών μελών. Να το συζητήσουμε κι άλλο. Πάντως βρήκα πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας. Σχετικά με πολλά από τα σχόλια του ΜΑΤ της Ενωτικής Αριστεράς. Συμφώνησα με πολλά από όσα λέτε. Είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια, πράγματι. Τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η έκθεση δεν περιλαμβάνει τα κατώτατα και ανώτατα όρια των φορολογικών συντελεστών. Κάτι που είπε ο κύριος Σάντ. Δεν υπάρχει διατύπωση μέσα στο κείμενο της εκθέσεως που προτείνει ελάχιστα ή ανώτατα όρια φορολογικών συντελεστών και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό απασχολεί πολλούς συναδέλφους και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να εμπλακούν και οι μικρές πολιτικές ομάδες όσο γίνεται περισσότερο και αναφέρομαι σε ορισμένα από τα σχόλια της μόλι από τους πράσινους. Ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τροπολογιών έγινε πολύ τεχνική πια η διαδικασία και η γραμματεία της Επιτροπής μας προσπαθεί να βάλει κάποια τάξη και να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια θέση όπου θα μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες, χωρίς όμως αυτές να οδηγήσουν πια σε ψεύδο συνενέσεις. Θέλουμε να περιληφθούν πράγματι όσο γίνεται περισσότερες πολιτικές ομάδες το, στην προσπάθεια δηλαδή. Τώρα για τις ε, λογιστικές επιχειρήσεις, accountancy firms, που είπε η Μόλι πάλι. Το συζητούμε αυτό με τον εισηγητή, θα το δούμε ξανά με τους σκιώδης ηγητές, ίσω μάλιστα να φτάσουμε και στην Ολομέλεια για να το συζητήσουμε αυτό, διότι βεβαίω υπάρχουν ποικίλε πολιτικέ απόψει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση επιχειρήσεων, βλέπετε τι είπε ο κ. Ζάνη, και αυτό είναι ζήτημα που απασχολεί του σιγητές και σκιώδη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί για την ώρα μία προσέγγιση των δύο βημάτων για να τεθεί σε ισχύ αυτός, αυτή η βάση CCCTB. Ίσως πρέπει να επιταχύνουμε. Αυτή είναι η δική μας γνώμη. Θα δούμε πώς θα το περιγράψουμε. Σε ό,τι αφορά τους καταγγέλλοντες. Το κείμενο είναι χρήσιμο. Σε ορισμένε περιπτώσει, βέβαια, υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει και που μιλούμε για ένα ταμείο για την υποστήριξη των καταγγελόντων. Το θέμα τώρα για <clears throat> την διαφάνεια, θέμα που έθιξε πάλι ο κύριος Ζάνη, ερχόμαστε στο κείμενο της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας και αυτό μπορεί να βοηθήσει όντως και ορισμένοι εξημών που έχουμε διαβάσει τα έγγραφα αυτής της Επιτροπής νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσουν. Θα χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες και για το Μητρό Εγγραφής Επιχειρήσεων και τα άλλα σχετικά. Το ζήτημα για το ρόλο των τραπεζών. Μέρος του κειμένου έχει υποβληθεί και σε μια προσπάθεια αντιμετώπιση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Τέλος, οι τελευταίοι δύο μιλητές, Φερνάντες και Σαντ, συμφωνώ με τα όσα είπατε για τους φορολογικούς παραδείσους, κύριε Φερνάντες. Έχουν κατατεθεί οι σχετικές διατυπώσεις και τα κριτήρια για τον καθορισμό των φορολογικών παραδείσων, για τον χαρακτηρισμό καλύτερα. Και το βασικό εδώ είναι ότι πρέπει να υπερβούμε τα όρια της προσέγγισης του ΟΟΣΑ. Τέλος, για κάτι που είπε ο κ. Όπως είναι τώρα η έκθεση, είναι ήδη διαρθρωμένη σε τρία τμήματα. Παραρτήματα, συστάσεις, διαφάνεια, συντονισμός, σύγκληση. Σε ό,τι αφορά την σύγκληση, η έκθεση μας δεν τοποθετείται σε ό,τι αφορά ανώτατα και κατώτατα όρια φορολογικών συντελεστών. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σύγκληση διαδικασιών, συστημάτων και ορισμών. ώστε να γίνεται ο ανταγωνισμός έντιμα και καθαρά και όχι από την πίσω πόρτα. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα μπορέσουν να εξετάσουν το θέμα υπό αυτό το πρίσμα και να τα δεχτούν. Σας ευχαριστώ πάντως όλες και όλους για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ Ανελίζ. Προβλέπετε η ψηφοφορία και ελπίζω έως τότε να είναι ε, ε, επιτυχής η διαπραγματεύσεις σας για την 1η Δεκεμβρίου. Για την Ολομέλεια προβλέπουμε τον Ιανουάριο. Ακούω όμως ότι και οι δύο εισηγητές ενδιαφέρεστε να το προτάξετε, δηλαδή να το βάλετε ήδη τον Δεκέμβριο. Άρα θα πρέπει να ε, κλείσουμε την 1η Δεκεμβρίου για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών. Αλλιώ δεν ε, προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν οι διάφορες πολιτικές ομάδες θα κάνουν την προσπάθεια να ε, προχωρήσουν. Έληξε αυτό το σημείο και έτσι φτάνουμε στο επόμενο. Η Σιλβί Γκουλάρ είναι έτοιμη, σωστά, για το σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων. Με συγκίτρια την κυρία Σιλβί Γκουλάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ε, τιμή σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους. Α, θα μιλήσω γαλλικά, μια που έχουμε καλούς διερμηνείς. Δεν χρειάζεται να μιλήσω αγγλικά, λέει η κυρία Κούλαρ, περνώντας από τα αγγλικά στα γαλλικά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Έβαλε και ο πρόεδρος τα ακουστικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους Σκιώδης και όλους τους υπόλοιπους. 177 τροπολογίες έχουμε. Θέλουμε να οργανώσουμε διάφορες συναντήσεις με τους σκιώδες. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε μια τέτοια συνάντηση πριν προχωρήσουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Έχω τέσσερις παρατηρήσεις και ένα συμπέρασμα. Πρώτη παρατήρηση. Από τότε που έκλεισε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, παρουσίασε ένα νομοθετικό κείμενο βάσει του άρθρου 138 της συνθήκης για την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Δηλαδή με τον έναν τον άλλο τρόπο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Κάποιες τροπολογίες έτσι κι αλλιώς ήταν είτε υπέρ είτε κατά της μνήας που γίνεται στην έκθεσή μου που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει για αυτήν την ενιαία εκπροσώπηση. Οπότε θα δούμε τώρα αν συμφωνούμε οι σκιώδες εισηγητές ή όχι. Το λέω για να το έχετε ακούσει όλοι, να το ξέρετε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δουλέψει και εμείς πρέπει να δούμε πού συμφωνούμε και πού όχι. Δεύτερον, θα συγκεντρώσω τροπολογίες διάφορες υπό τον τίτλο «Διαφάνεια». Διάφορες προτάσεις έχουν γίνει από τους συναδέρφους με διαφορετικούς βαθμούς ε, λεπτομέρειες. Ο κύριος Γκίκολ προσπάθησε να πάει πιο μακριά. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Αλλά μετά πρέπει να δούμε τι είναι προτιμότερο να κάνουμε, τι είναι ρεαλιστικό. Πόσο μακριά δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια έκθεση πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου μα. Πρέπει να πάμε σε λεπτομέρειε, πρέπει να θέσουμε αρχέ. Θα το συζητήσουμε μεταξύ μα. Πάντω υπάρχει συμφωνία. Κάποιε τροπολογίε επιμένουν στο γεγονό ότι κάποιοι οργανισμοί δεν δίνουν αρκετό χώρο στο θέμα της διαφάνειας απέναντι στους καταναλωτές, το θέμα των ε, μισθωτών. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, μπορεί να είναι μια καλή διευκρίνηση, αλλά θα δούμε πώς θα συμπεριληφθεί στο κείμενο. Θέλω επίσης να τονίσω ότι ο κύριος Δράγκη, όταν ήρθε την τελευταία φορά στην Επιτροπή μας και τον ρώτησα κάτι, έδειξε να δέχεται ένα άνοιγμα όσον αφορά την διαφάνεια για τις θέσεις που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τους συνεργάτες στην ΕΚΤ να δουλέψουμε για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα χωρίς μεγάλες αλλαγές. Γιατί αν υπάρχει βούληση από πλευρά των θεσμικών οργάνων, τότε έχουμε κερδίσει. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να χτίσουμε είτε επισημοποιήσουμε αργότερα με θεσμική συμφωνία τα πράγματα είτε όχι. Τρίτον, για το θέμα accountability της λογοδοσίας. Ίσως χρειάζονται πιο συγκεκριμένες προτάσεις από ό,τι είχαμε στην πρώτη έκθεση. Νομίζω ότι και εδώ υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το ότι πρέπει να βελτιωθεί η λογοδοσία. Δηλαδή όταν πρόκειται για την Επιτροπή, άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα κλπ. Είτε πρόκειται για την ΙΟΠΑ, για την ΕΣΜΑ, για την Ευρωπαϊκή και την ε, Τράπεζα Επενδύσεων κλπ. Και για άλλα όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια, καλό είναι να ενισχυθεί ο διάλογος μαζί τους, να διαρθρωθεί καλύτερα, να δομηθεί καλύτερα και με ρεαλισμό και μάλιστα με την προοπτική επισημοποίησης ίσως των επαφών αυτών και του διαλόγου. Τέταρτο σημείο. Τι κάνουμε με τις θέσεις των χωρών μελών στα διάφορα όργανα. Είτε πρόκειται για τους G20, είτε πρόκειται για άλλα όργανα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μιλάει, της μία που εκπροσωπείται και εκείνη και κάποιες χώρες μέλη όταν σε συναπόφαση υιοθετούνται κάποια μέτρα και που δεσμεύονται και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αλλιώ από άλλε περιπτώσει. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει κάτι για να προχωρήσουμε βάσει των όσων έχουν κερδιθεί μέχρι τώρα. Α πούμε με την Τραπεζική Ένωση. Οι χώρες μέλη δέχτηκαν την πρόοδο για την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε καταλήξει σε κοινή νομοθεσία, έχουμε καταλήξει σε κοινά όργανα. Τώρα, είτε πρόκειται για την EBA, είτε πρόκειται για την ε, αρχή τραπεζών δηλαδή, είτε πρόκειται για κάτι άλλο, πρέπει να υπάρχει συνοχή. Ήμουνα στην Ουάσιγκτον τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και εκεί συναντήθηκα με διάφορους εταίρους εν ώψη της έκθεσης αυτής και με εντυπωσίασε η σύγκληση εδώ δεν λέω ότι στην Αμερική η σύγκληση είναι τέλεια, εννοείται ότι δεν συμφωνούμε με διάφορα σημεία, αλλά οι Αμερικανοί εταίροι θέλουν να υπάρχει αυτή η σύγκληση στην Ευρώπη. Μίλησα με τον γερουσιαστή Σέλβι που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής που ασχολείται με τα τραπεζικά ζητήματα εκεί. Στο Κογκρέσο λοιπόν έχουμε την αίσθηση ότι αναρωτιούνται τέτοια πράγματα για τη λογοδοσία, για το πώς ε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε με εμπειρογνώμονες, αλλά τα δημοκρατικά όργανα θα εξακολουθούν να έχουν εκείνα την ευθύνη για την ομοθέσια. Και στην Αμερική υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που καθορίζουν προσανατολισμούς και άλλα, όπως το κείμενο του Φρανκ, αλλά υπάρχει ιδέα αυτή του συντονισμού Υπάρχει ένας κοινό προσανατολισμός. Ξέρετε ότι τα οικονομικά δεν βρίσκονται μέσα στο TTIP, ξέρετε ότι τα benchmarks και άλλα δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, αλλά ίσως είναι ευκαιρία η ατζέντα αυτή να προχωρήσει και διατλαντικά, χωρίς αποκλεισμούς, για να προχωρήσουμε στις δύο ζώνες που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ε, χρηματοοικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίω. Συμπέρασμα να υιοθετήσουμε αυτό που προτείνει λίγο πολύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι η κοινή λογική. Δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ρεαλιστικά, χωρίς να βάζουμε ιδιαίτερα επίμαχα ζητήματα, αλλά να βοηθούμε τους εταίρους να συμπορευτούν μαζί μας. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στο Συμβούλιο που θέλουν να ενισχύσουν το συντονισμό και για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον να ξέρουμε ότι οι αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρώπη πρέπει να μπορούν να στηριχτούν και να προωθηθούν και διεθνώς. Οπότε πώς θα αποφύγουμε κάποιες χώρες μέλη σε διεθνή φόρα τελικά να αντιμάχονται αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε αυτό που έχουμε αποφασίσει εδώ μέσα στην Ευρώπη και αυτό το οποίο εκπροσωπούμε στο εξωτερικό. Είτε πρόκειται για την Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία κυρίως αυτή επηρεάζεται από τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτή είναι η γενική μου προσανατολισμή. Δεν θέλω να προκαθορίσω τι θα αποφασίσουμε τελικά με τους σκιώδεις, πάντως πιστεύω ότι θα βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Θέλω να συνεργαστώ με όλες τις πολιτικές ομάδες και θέλω ευρύτατη συνένεση. Εννοείται ότι υπάρχουν τροπολογίε όπου φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει η κοινή ευρωπαϊκή θέση σε διεθνή φόρα. Δικαιωμά Αλλά τέτοιε τροπολογίε ίσω δεν θα συμπεριληφθούν την τελική συμφωνία που θα πηγαίνει μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση. Περιμένω τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Σιλβί και συνεχίζουμε με την Σύρπα που είναι σκιώδη συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ την Σιλβί για την θαυμάσια συνεργασία. Πραγματικά ε, θαυμάσεις διανοητικές ικανότητες και πολλή δουλειά. Και το δείχνει αυτό και με τις αναλύσεις που κάνει στις τροπολογίες. Ο χωρισμός σε τέσσερις κατηγορίες πολύ καλά έγινε, δηλαδή περιλαμβάνει τα θέματα που συζητούμε Τα ταξινομεί και τις τροπολογίες και νομίζω κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Σας άκουσα να λέτε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η αύξηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της ε, συνοχής στην δράση. Και φαίνεται να υπάρχει συμφωνία επ' αυτών. Τα άλλα θέματα βέβαια είναι πόσο τολμηρός θα φανεί κανείς ή πόσο τολμηροί θα φανούμε και για το θέμα της ε, ενίας έδρας. Εδώ στο Κοινοβούλιο ωστόσο εδώ σημειώνεται πολιτική διάσταση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε εδώ μεταξύ μας ποια γραμμή θα κρατήσουμε. Εγώ φοβούμαι προσωπικά ότι κινούμεθα υπερβολικά προσεκτικά, δηλαδή λέμε κάτι για τα πάντα και για την ισορροπία μεταξύ χωρών μελών και των αρμοδιοτήτων χωρών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι τελικά από τόσο, να είμαστε τόσο πολύ προσεκτικοί δεν προχωρούμε πολύ. Προτιμώ να είμαστε λίγο πιο τολμηροί και να λάβουμε υπόψη τις δυνατότητες που μας ανοίγονται με τις τροπολογίες, γιατί αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, αλλά και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την θέση των ε, επιχειρήσεών μας ανά τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι έλασον θέμα αυτό, δεν είναι καμιά ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το ποια είναι η θέση της Ένωσης. Είναι σημαντικό, είναι μείζον θέμα πώς θα διαχειριστούμε την ανταγωνιστικότητά μας, την ανάπτυξή μας και ποια είναι η θέση μας στον κόσμο σε όλα αυτά και πώς φτιάχνουμε καλύτερη νομοθεσία. και ποια πράγματα απασχολούν τους εταίρους μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και επίσης σας ενθαρρύνω να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Και αυτή η προπολιτική επιχειρηματολογία, η, ο προβληματισμός. Για παράδειγμα για το shadow banking θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε να πούμε κάτι ως πολιτική. Και για το crowdfunding που αρέσει σε όλους μας, σε όλες και όλους μας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εάν δεν υπάρχει μια αναλογική νομοθεσία κάποιος θα την πατήσει και πολύ άσχημα, πολύ σύντομα. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα πολιτικά να το προωθήσουμε και όχι μόνο με στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Και ένα άλλο θέμα, πιο τεχνικό. Η σύσταση BEPS του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, θα, του δηλαδή, θα πούμε τα ίδια πράγματα όπως το FRS σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δηλαδή θα υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στα διάφορα μέρη του κόσμου, ε, δημιουργώντας έτσι επικαλύψεις. Άρα πιο ενωτική, πιο συνεκτική γραμμή, βεβαίως πρόκειται για θέμα ανταγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να λάβουμε υπόψη τους κανονισμούς αλλά και για την σύνταξη προδιαγραφών γιατί και εδώ δημιουργούνται προηγούμενα Και όλα αυτά και για την οικονομική πολιτική ε, γενικότερα που είναι η οικονομική πολιτική άλλη υπόθεση. Ε, εκεί βέβαια η διαφάνεια είναι πρώτη προτεραιότητα. Thank you very much, Sirpa. For the S&D group, I give the floor to Ευχαριστώ. Μάτι Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να τα πω στα γαλλικά. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Γκουλάρ και να την συγχαρώ βέβαια για την εκθεσή της και να την ευχαριστήσω για την ε, προσέγγιση της που ήταν ε, ε, τέτοια που μας συμπεριέλαβε όλους. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στα όργανα και ιδίω στις χώρες μέλη είναι ότι θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, accountability δηλαδή, λήψη υπόψη του γενικού συμφέροντος, του, του γενικού συμφέροντος, της ε, δημοκρατίας και, ναι, και Και είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό να ε, ληφθεί υπόψη, μάλλον να, να γίνει δεχτό από μια μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβουλίο μας. Βλέπουμε μια σύγκληση για τον ρόλο του Κοινοβουλίου, για την ε, δημοκρατία, το ε, δημόσιο συμφέρον, τη λογοδοσία. Ε, για τη διαφάνεια αρχίζουν οι αποχρώσεις. Είμαστε υπέρ ενό υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας. Εδώ όμως θέλω να προσθέσω ότι ωραία είναι η διαφάνεια, αλλά υπάρχει κίνδυνος να πνίξουμε με υπερβολικά δεδομένα και πληροφορίες τους καταναλωτές και πολίτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει και μια τεχνογνωσία από την πλευρά των καταναλωτών, των πολιτών, γι' αυτό να υποστηρίξουμε τις ε, μη κρατικέ οργανώσεις που δρούν προς το συμφέρον των καταναλωτών και των πολιτών γενικότερα. Όσον αφορά την εκπροσώπηση στην ε, Eurogroup και στη ζώνη ευρώ, δεν υπάρχουν και αποκλήσει. Η δική μας πολιτική ομάδα θέλουν μια ενιαία εκπροσώπηση του Eurogroup και της Ένωσης. Αυτό δεν θα γίνει βέβαια αμέσω, θα χρειαστούν μικρά βήματα, αλλά σταθερά. Χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση και χρειάζεται και μια προοπτική. Άρα, χρειάζεται κάποια ημερομηνία για να υπάρξει αυτή η ενιαία ε, εκπροσώπηση. Ίσως αυτό να, το στοιχείο να προσφέρει και μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην πρόταση. Εγώ νομίζω ότι η Ένωση δεν είναι υποχρεωμένη να μιλεί με μια φωνή. Αλλά αυτό που θα λέει και όσοι φωνές και να μιλούν για λογαριασμό της θα πρέπει να δίνουν το ίδιο μήνυμα. Γιατί βαρύνει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Εδώ με εκπλήσει κάτι. Θεωρεί κανείς πραγματικά ότι μια χώρα μέλος όσο σημαντική και αν είναι στα πλαίσια της Ένωσης ότι μπορεί να σταθεί μόνη της απέναντι στις ΗΠΑ, στην Κίνα ή άλλους γίγαντες της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Είναι λίγο δημαγωγικό να προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι η σωτηρία τους βρίσκεται μόνο στην προστασία των εθνικών συμφερόντων. Αυτά είναι ξεπερασμένες ε, θέσεις, ε, απερχιωμένες και δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σήμερων σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στα, στο παγκόσμιο αυτό οικονομικό γίγνεσθε, χρειάζεται κοινή δράση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, να στηρίξουμε την ένωση, το νόμισμά μας και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν χαίρομαι που βλέπω τροπολογίες από άλλες πολιτικές ομάδες που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση που ζητούμε να μην ε, γίνεται προσφυγή ε, ε, σε ιδιώτες, ιδιώτες διαιτητές, αλλά να υπάρχουν άλλα συστήματα και βέβαια να υπάρχουν και διασυνδέσεις με το χρηματοοικονομικό τομέα και έχουμε εκθέσεις, έχουμε κείμενα καλά θεμελιωμένα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τη συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Ο πρόεδρος Φέρμπερ, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την Ενωτική Αριστερά. Μιγέλ Βιέγας. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ε, ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν ε, συμφωνούμε με το περιεχόμενο, την ανάλυση και με μεγάλο μέρος ε, αυτής της έκθεσης. Για ξεκάθαρους και σαφείς λόγους. Ότι δηλαδή εμείς πολιτικώς είμαστε τοποθετημένοι στον αντίποδα όλου του πολιτικού ιδεολογικού υποβάθρου στο οποίο δράζεται αυτή η έκθεση. Κατανοούμε την ανάγκη σταθερότητας του οικονομικού συστήματος, γιατί αυτό εγγυάται την καλή χρήση και την κατανομή αυτών. Εκεί όμως που εμείς αποκλίνουμε είναι στη ρίζα, στην προέλευση της αστάθειας και της έλλειψης ε, ε, σταθερότητας και στους μηχανισμούς που προτείνονται για να διορθωθεί ή να ελεγχθεί η αστάθεια του οικονομικού συστήματος. Η αστάθεια αυτή, κατά τη γνώμη μας, ε, εκπορεύεται από την ιδιωτικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που ξεκίνησε το 1980 και η λύση περνά από τον τον κρατικό έλεγχο του ε, οικονομικού συστήματος και ζητώ συγγνώμη από τα ευαίσθητα ότα, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Ο, ο, ο χρόνος θα δείξει ότι έχουμε δίκιο. Πάντως, ε, όπως σας είπα, συμφωνούμε ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, συμφωνούμε ότι χρειάζεται περισσότερη θεμητότητα δημοκρατική των ε, θεσμών που μιλούν εξ ονόματος των λαών, συμφωνούμε με την ανάγκη να υπάρχουν και παγκόσμιοι κανόνες ε, στα θέματα διαφάνειας και ευθύνης των οργανισμών και του διαλόγου με τα πολιτικά όργανα, αλλά δεν συμφωνούμε με την ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, να μιλάμε ε, με μια μόνη φωνή ή που, όπως υπόθηκε εδώ με εντυπωσιακό τρόπο, είναι 28 χώρες που, το, που λένε το ίδιο πράγμα κατά βάση. Έτσι είπε κάποιος εδώ. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την ιδέα ενό παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, γιατί αυτό φυσικά απομακρύνει τα κέντρα λήψης αποφάσεων από τους πληθυσμούς. Όσο και αν προσπαθούμε εδώ να βάλουμε διάφορα μέτρα και ρήτρες και μηχανισμούς που υποτίθεται ότι θα συνδέουν και θα ε, νομιμοποιούν δημοκρατικά όλα αυτά τα κέντρα. Γιατί στην πράξη ξέρουμε πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτή η ιδέα είναι απολύτως ασύμβατη με την πολιτιστική, πολιτική, ιδεολογική πολυμορφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία δηλαδή ακολουθεί τη λογική μια, της ενιαίας σκέψης. Λες και υπάρχει μόνο ένα οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο ανάπτυξης και αυτό κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Δεν μπορεί να αρθεί η δυνατότητα και η νομιμότητα της κάθε χώρας να επιθυμεί να κατευθυνθεί προς άλλη, προς άλλη κατεύθυνση, άλλη πορεία. Ναι, μια φωνή, αλλά ποια φωνή θα είναι αυτή. Και αυτή τη φωνή που ακούγεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα συμφέροντα της, ε, των μεγάλων ε, χρηματοπιστωτικών ομήλων. Και γι' αυτό και έχουμε τόσες επιφυλάξεις. Και θέλουμε μάλιστα να δημιουργήσουμε εδώ ένα θεσμό που θα αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα φόρα. Ακόμα μια φωνή ώστε να μπορέσει να πει ξανά τα ίδια τροπάρια των ε, νέο φιλελεύθερων ε, θέσεων. Έχουμε κουραστεί από αυτό το πράγμα. Ακόμα ένα θεσμό δεν πρόκειται να προσθέσει κάτι ε, σε σχέση με τα αυτά που ήδη υπάρχουν και στη σημερινή πραγματικότητα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς στην Πορτογαλία Τώρα ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια συγκυβέρνηση που ονομάζεται της αριστεράς και συγκεντρώνει διάφορα κόμματα ε, από το αριστερό ιδεολογικό φάσμα. Και αυτό ε, μέσα σε ένα πλαίσιο ιδιωτικοποίησης δημόσιων οργανισμών μεταφορών που συνεχίζεται στη δημόσιο τομέα. Αυτό είναι τελείως αντίθετο με τις συστάσεις που μας, επιβλήθηκαν από το εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Ασυμβατότητα μιας μοναδικής πολιτικής και ιδεολογικής κατεύθυνσης που τελικά δεν συμφωνεί με τις ε, ε, διεκδικήσεις των λαών, όπως φάνηκε από τις τελευταίες εκλογές, όπου φάνηκε δηλαδή ότι ο πορτογαλικός λαός ζητά μια βαθιά ε, τομή, μια βαθιά αλλαγή σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείται μέχρι στιγμή στη χώρα μας. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι δεν χρειάζεται ακόμα ένα μέσο που θα ε, αλλοιώσει την κυριαρχία των λαών, των κρατών και του πορτογαλικού κράτους στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας ενός ε, προγράμματος με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. I think that is... Βέβαια, αυτό ξεπερνάει τα όσα συζητάμε τώρα, αλλά η Σιλβή εντάξει, τα ακούει. Εκ μέρους των Πρασίνων. Θα δικαστείτε το Σβέν. Ναι, ναι, εξακολουθώ να είμαι ο Σβέν. Ωραία, Σβέν. Πες μας μέσω του Φίλιπ Λαμπέρτε; Για σήμερα όμω, μόνο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ε, Σβέν για πάντα, είναι ένα αντικατάστατο εννοείται. Ναι. Δεν χρειάζεται να μιλάω εκ μέρου κάποιου άλλου. πάντων, θα αρχίσω γαλλικά, αλλά επειδή σημειώσουμε στα αγγλικά, του Σβέν δηλαδή, θα το γυρίσω στα αγγλικά μετά. Λοιπόν, η πράσινη είμαστε πιο πολύ πέρα της προοπτικής μιας ε, όσο γίνεται πιο ενωπημένης ε, Ευρώπης, ομοσπονδιακής. Γι' αυτό και συμφωνούμε με το πνεύμα της εισηγήτριας. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Όμως, αυτή η όλο και πιο στενή ολοκλήρωση δεν είναι δυνατόν να οδηγεί σε μείωση της ποιότητας της δημοκρατίας ουσιαστικά των καθεστώτων μας. Και ξέρω ότι συμφωνεί και η Σιλβή. Διαπιστώνουμε όμως ότι συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή ότι με την κρίση του ευρώ βλέπουμε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό επίπεδο συνοδεύεται από μια ονομαστική αδυναμία του δημοκρατικού ελέγχου. Και γιατί τον λέω ονομαστικό, γιατί δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει για την ποιότητα δημοκρατικού έλεγχου που ασκείται σε εθνικό επίπεδο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση για παράδειγμα, θα ήθελα δηλαδή ειλικρινά όλα τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν έναν ρόλο δημοκρατικού ελέγχου όπως έχει σήμερα η Μπούτουσταξ στην Γερμανία. Που αποτελεί παράδειγμα που δεν ακολουθούμε συχνά στην Ευρώπη. Θα σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Στη Bundestag, αν οι βουλευτές θέλουν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα της κυβέρνησης, έχουν το δικαίωμα να έχουν αυτή την πρόσβαση. Σε πολλές χώρες μέλη, στη δικιά σου, στη δικιά μου, δίνουν αγώνα οι βουλευτές προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικά έγγραφα. Απίστευτο. Άρα μην βλέπουμε τα πράγματα άσπρο μαύρο μη λέμε ότι όσα γίνονται σε εθνικό επίπεδο είναι καλά και όσα γίνονται στην Ευρώπη δεν είναι. Όχι, γιατί υπάρχουν πολλέ αποχρώσεις του γκρι ανάμεσα στα δύο. Υπάρχει θέμα δηλαδή εδώ και δεν είναι μόνο θέμα διαφάνεια, Μια λέξη που εμένα δεν μου αρέσει και τόσο πολύ, αλλά πάντως στα γαλλικά εσείς είπατε accountability. Γιατί, γιατί στα γαλλικά δεν έχουμε την κατάλληλη λέξη για να απεικονίσουμε αυτό που σημαίνει στα αγγλικά accountability αυτή τη λογοδοσία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε έχει να κάνει με αυτό ακριβώς και μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι όταν πρόκειται για την Ευρωζώνη. Πολλά μένει ακόμα να γίνουν και κυρίως να ενισχύσουμε το κομμάτι αυτό του κειμένου, που εντάξει καλό είναι, αλλά να ζητήσουμε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να προβλέψουν διοργανική συμφωνία για να επισημοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο δίνεται εντολή στην Επιτροπή όταν αυτή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωζώνη σε διεθνή φόρα. Μια συγκεκριμένη περίπτωση που θέλουμε εδώ να θίξουμε είναι τον ΙΣΒ, που καθορίζει τα λογιστικά πρότυπα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Και παρόλο που σήμερα λειτουργεί με αδιαφανή τρόπο, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποφεληθούμε από την έκθεση αυτή προκειμένου να πούμε ότι Πρέπει να προσέξουμε πολύ καλύτερα τι γίνεται και τα ευρωπαϊκά όργανα να είναι εκείνα τα οποία δίνουν την όθηση για τα λογιστικά πρότυπα. Θέλω επίσης να επαναλάβω και κάτι άλλο με το οποίο είχαμε συμφωνήσει με μεγάλη πλειοψηφία όταν είχαμε την έκθεση για την Τρόικα. Πρόκειται για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Όταν συζητήσαμε την έκθεση εκείνη, είχαμε συμφωνήσει για την αναγκαιότητα να έχουμε έναν διεθνή μηχανισμό αναδιάρθρωσης των ε, χρεών των χωρών μελών. Η έκθεση μιλάει βέβαια για ε, οργανισμούς και όχι για το περιεχόμενο. και κάτι για να δώσω μια απόχρωση στην προσέγγιση αυτή την ομοσπονδιακή για την οποία σας μίλησα πριν. Σήμερα στην κατανομή αρμοδιοτήτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια για τα πάντα. Ακόμα και σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Αν λοιπόν θέλουμε το μήνυμά μας να είναι ισχυρό, πρέπει να δούμε πώς διατυπώνουμε τα πράγματα, πώς τα εκφράζουμε, ώστε μέσω αυτής της ενιαίας εκπροσώπησης προσοχή να μην ε, εποφελείται από αρμοδιότητες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει και έχουν οι χώρες μέλη. Τότε δεν χρειάζεται να υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση, αλλού όμως εκεί όπου έχει οι αρμοδιότητες προφανώς και πρέπει να είναι κοινή η εκπροσώπηση και ενιαία. Αυτά είχα να πω και φυσικά ο Σβέν δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα υποστηρίξει τις θέσεις μας ε, με μπρίο. Τελικά τα από όλα στα γαλλικά. Δεν μίλησα αγγλικά. Πρόεδρος. Η ευθυντή Μαρκοτσάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της. Εγώ θα μιλήσω για τα δύο θέματα που υπάρχουν περισσότερες διαφορές σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Καταρχήν, πριν να μιλήσω για τις διαφορές, να πω αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Και αυτό με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα, που είναι δύο βασικά θέματα στο πλαίσιο αυτή της ε, έκθεσης. Για τη διαφάνεια, για τη διαφάνεια πούμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο σύνολο των ομάδων και στο σύνολο τη ομάδα εργασία. Είναι απαραίτητο όντω αυτοί οι οργανισμοί που έχουν παίξει τόσο σημαντικό ρόλο και εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο τη διαχείριση τη κρίση και του χρηματοπιστωτικού συστήματο, να μπορούν να έχουν να είναι πραγματικά διαφανείς και αυτό είναι κατανοητό και για τους ίδιους τους πολίτες που συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τη λογική ή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτούς τους οργανισμούς. Και έπειτα ε, κάτι ακόμα ε, επί το συμφωνούμε είναι ο δημοκρατικός ε, έλεγχος επί το οποίο οι συνάδελφοι εξέφρασαν τη γνώμη τους γιατί πιστεύω ότι υπό αυτή την άποψη είναι απαραίτητο στην έκθεση αυτή να προσπαθήσουμε, να ζητήσουμε, ε, να απαιτήσουμε μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το μοναδικό όργανο άμεσα εκλεγμένο από τους ε, ψηφοφόρους να έχει μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ένωση στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών. Ε, τόσο στο στη φάση του ορισμού, όσο και στη φάση του ελέγχου για το ποιες αποφάσεις ελήφθησαν. Αυτά είναι τα οποία υποστηρίζουμε και που ε, ελπίζω πως θα καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικές και σε ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου. Το τμήμα για το οποίο συμφωνούμε λιγότερο και φαίνεται και από τις τροπολογίες μας είναι το τμήμα που αφορά την ενιαία εκπροσώπηση της Ένωσης σε αυτούς τους οργανισμούς. Πιστεύω και βέβαια αυτή είναι μια τελείως πολιτική ε, θέση και οι θέσεις μας γι' αυτό και ενδιαφέρουν. Πάντως κάτι το αντικειμενικό, ένα αντικειμενικό στοιχείο είναι ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει πως δεν είναι σε θέση, δεν είναι έτοιμη να έχει μια ενιαία εκπροσώπηση και άρα το να προτείνουμε κάτι τέτοιο ε, ίσως να είναι τελικά αντιπαραγωγικό. Νομίζω όμως πως ε, τη σήμερον ημέρα είναι περισσότερο απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας σοβαρά τις διαφορές που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητο κάθε κράτος μέλος να μπορεί να προστατεύει τα χαρακτηριστικά του συστήματός του εντός των οργανισμών αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις που μπορεί να έχουν ε, πολύ σημαντικό αντίκτυπο επί των διαφόρων ε, ε, χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάμε σήμερα για την απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σύνολο δυνατότητας απορρόφλαψης, or capacity. Μιλάμε δηλαδή για τα μέσα απορρόφησης ε, της απώλειας κεφαλαίου, επιπλέον μέσα για τις τράπεζες που είναι συστημικές. Αυτό του είδους οι αποφάσεις λοιπόν ε, ζημιώνουν τις τράπεζες που έχουν περισσότερο θέση εμπορικών τραπεζών ε, και στο Ιταλικό σύστημα βασίζονται σε αυτό οι τράπεζες, ενώ δεν ζημιώνει, δεν τιμωρεί τις επενδυτικές τράπεζες που είναι πιο ε, επικίνδυνες. Το σύστημα δηλαδή βασίζεται περισσότερο τις ε, ε, εμπορικές τράπεζες, τις επενδυτικές τράπεζες και αυτό ε, είναι αγγλοσαξονική παράδοση και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα που σας δίνω ότι όχι, για το ότι υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες και ότι για το ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο αυτών των οργανισμών μπορεί να έχουν αντίκτυπο και αρνητικό αντίκτυπο πολύ διαφορετικό ανάλογα με το ποια είναι η δομή του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος που υπάρχει σε κάθε χώρα. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η συζήτηση που γίνεται σήμερα όχι μόνο στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών αλλά και στο εσωτερικό του Ευρωκοινοβουλίου για το πώς λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι, θεσμική η οι ελεύθερη κινδύνου, οι ελεύθερες κινδύνου επενδύσεις, οι τράπεζες οι οποίες μέσα στη χαρτοφυλάκια τους έχουν κρατικούς τίτλους. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Ένα παράδειγμα, εάν σήμερα αποφασίζαμε ας πούμε ότι οι κρατικοί τίτλοι ε, βεβαίως από τεχνικής άποψης και η κρίση το έχει αποδείξει δεν είναι μέσα μηδενικού κινδύνου, η κρίση το έχει αποδείξει αυτό, μπορούσαμε να ζητήσουμε δηλαδή μεγαλύτερη αξία. Ο αντίκτυπος στα διαφορετικά τραπεζικά συστήματα θα είναι τεράστιος. Οι Ιταλικές τράπεζες έχουν ε, στο χαρτοφυλάκια τους 400 ε, δις ευρώ ε, κρατικού ιταλικών ομολόγων και αυτό βέβαια λόγω πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν και υποχρέωσαν τις τράπεζες να αναλάβουν αυτά τα μέσα στους προπολογισμού τους. Επειδή έχουν τριπλό β μείον ή τριπλό β συν, μπορεί αυτοί οι τίτλοι να μειωθούν ε, κατά 40% και οι τράπεζες οι Ιταλικές να υποχρεωθούν να συλλέξουν 200 εκατομμύρια κεφάλαια επιπλέον. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές, όπως είπα, ευαισθησίες στο εσωτερικό αυτών των μηχανισμών και γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προστατέψουμε αυτές τις διαφορές. Ελπίζω πως θα υπάρξει η ευκαιρία, αν και ξέρω πως η θέση της εισηγήτριας αλλά και κάποιων μεγάλων ομάδων είναι να τίνουν και προς σταδιακά προς μια ενιαία εκπροσώπηση, ωστόσο ελπίζω πως θα, μεταξύ μας θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό για να ληφθούν υπόψη και αυτά τα προβλήματα που ανέφερα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον άλλον για την ώρα. Άλλη συνάδελφη. Α, να, κάποιος ακόμα ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Έχετε αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη χώρα μου, τη Ρουμανία, ήμουν μέλος της ε, Εποπτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων και στη συνέχεια της ε, Εποπτικής Χρηματοπιστωτικής Αρχής. Και λαμβάνοντας υπόψη και μελετώντας αυτή την έκθεση, θα ήθελα να πω ε, κάτι για τα ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα, ας πούμε αυτό που εποπτεύει τον ασφαλιστικό τομέα, αυτό που εποπτεύει το τομέα την ΕΣΜΑ, των ε, κινητών αξιών και, τα, και το ε, των ειδικών τραπεζών. Όλα αυτά συνδέονται με διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη γνώμη μου ε, επικρατεί χάος εάν λάβουμε υπόψη την εκπροσώπηση αυτών των θεσμών, των ευρωπαϊκών θεσμών σε διεθνές επίπεδο και σε διάφορα ε, ε, διεθνή σώματα. Έχουμε την ΕΣΜΑ, την ΕΙΟΠΑ και την EBA, ε, την Τραπεζική Αρχή. Όλα αυτά εποπτεύουν διάφορους τραπεζικούς τομείς Υπάρχουν και διάφοροι αντίστοιχοι διεθνείς οργανισμοί που ορισμένες φορές ωστόσο, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί οργανισμοί με εκπροσώπους τους στα διάφορα διεθνή σώματα. Υπάρχουν επικαλύψεις ε, στην εκπροσώπησή μας στα διεθνή φόρα. Ενώ ταυτόχρονα σε επίπεδο των κρατών μελών και η έκθεση Ευρωπαίων εκπροσώπων στις διεθνείς οργανισμούς για να ενσωματωθούν εκεί και να μπορέσουμε να έχουμε τα πρακτικά στοιχεία του πρακτικής οργάνωσης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στους διεθνείς οργανισμούς, καταρχήν θα, πιστεύω πως θα πρέπει να τυποποιηθούν πολύ καλά οι εθνικοί υποπτικοί ε, οργανισμοί των κρατών μελών. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι στις 28 ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν διαφορετικοί εποπτικοί οργανισμοί, ορισμένοι εκ των οποίων είναι ξεχωριστοί. Εποπτεύουν την ασφάλιση, τα, ε, τις αγορές ε, τίτλων κτλ. Και η εκπροσώπηση τους σε επίπεδο στην ΕΣΜΑ, στην ΕΙΟΠΑ και στην EBA είναι τελείως διαφορετική. Πρέπει δηλαδή να τυποποιήσουμε εάν θέλουμε να έχουμε κοινή, κοινά εποπτικά ευρωπαϊκά όργανα και να μπορούν ε, εύκολα και να, να ε, λειτουργήσουν και να έχουν αποτελέσματα. Πρέπει να καλέσουμε τα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να υπάρχουν ένα, δύο, τρία διαφορετικά σώματα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί Ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιποποιηθεί και η εκπροσώπηση των ε, ευρωπαϊκών ε, μας οργάνων στα διεθνή όργανα. Δεν είναι ούτε και ξεκαθαρά τα πράγματα, υπάρχουν επικαλύψεις Υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί για τις δεξιδοτικά ταμεία, για τις ασφαλίσεις κτλ. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε για το επόμενο στάδιο. Για τη χώρα μου, τη Ρουμανία, το 2013 οι τρεις εποπτικές αρχές συγχωνεύθηκαν μέσα σε 24 ώρες. Αλλά τώρα λειτουργούν ως ένα σώμα, ως μια αρχή για την εποπτεία των τριών αυτών αγορών. Ενώ υπάρχουν τρεις αντιπρόεδροι. Ωστόσο δεν υπάρχουν ε, συνεργασίες ανάμεσα των τριών σκελών ας πούμε του ίδιου οργανισμού. Ένας πρόεδρος, τρεις αντιπρόεδροι και συνεδριάζουν μόνο σε επίπεδο συμβουλίου. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Πρέπει να ε, οργανωθούμε καλύτερα, ώστε να εκπροσωπούνται οι χώρες μας και καλύτερα στη Φραγκφούρτη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Φερνάντες, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο Γουλάρ για την έκθεσή της. Πιστεύω πως ε, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην ε, ευρωπαϊκοποίηση και την ομοσπονδιοποίηση της Ευρωζώνης. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ε, εκθέσεις. Η έκθεση των πέντε προέδρων επίσης ενσωματώνει αυτή την ενοποίηση, ενοποίηση για την οποία χαίρομαι, ενώ ταυτόχρονα όμως χαίρομαι, λυπούμε γιατί η έκθεση των πέντε προέδρων ε, δεν μιλά παρά για την εκπροσώπηση της Ευρωζώνης από τον ε, πρόεδρο του Ευρωγκρουπ. Ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η εκπροσώπηση αυτή να γίνεται από το εκτελεστικό σκέλος, το όργανο της ε, Ένωσης. Άρα λοιπόν να είναι επίτροπος ε, οικονομίας που θα πρέπει να δίνει την γνώμη όλων, δεν μπορεί να δίνει οποιαδήποτε κομματική προσωπική θέση. Πάντως η ευθύνη θα πρέπει να επιβαρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το Eurogroup. Εν πάση περιπτώσει, εκπροσώπηση στο διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, στη Διεθνή Τράπεζα ή στις διάφορες αναπτυξιακές τράπεζες, όπου πιθανότατα θα πρέπει να ε, προωθήσουμε αυτή την ενοποίηση και σίγουρα η πιθανότητα θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την εννοποίηση. οπου πιθανοτατα θα Τράπεζα και σιγουρα η διεθνη τραπεζα ειναι η πιο σημαντική σημαντική γιατί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν δικαιολογείται εύκολα. Είναι μια ευκαιρία το Ευρωκοινοβούλιο να έχει μια ξεκάθαρη φωνή και είμαι βέβαιος πως θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος Φέρβερ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο επειδή έχω καταθέσει μια από τις ε, προτάσεις, έχει νόημα το ερώτημα εάν δεν πρέπει να ξεχωριστούν η κεφαλαιακή κατάθεση από την ευθύνη. Ίσως να διαχωριστούν αυτά. Αν είναι δυνατόν η η συγγετρία να πει κάτι. Έχει το λόγο, ε, κυρία Γκουλάρ. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ευχαριστώ σαν θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, γνωμοδοτήσει. Κανονικά το λόγο τον δίνει βέβαια ο Πρόεδρος, αλλά αν πάντως ε, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ. Μα θα είμαι συντομότατη κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ του εγγράφου εργασίας και της σημερινή συζητήσεω η Επιτροπή έχει καταθέσει κείμενο για την προς τα έξω εκπροσώπηση. Διαβάζοντας την έκθεση και τις περισσότερες τροπολογίες βρίσκω ότι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε την πρόταση ως μέρος της εφαρμογής της εκθέσεως των πέντε πρόεδρων. Προ τα έξω εκπροσώπηση δηλαδή, να σημαίνει ότι μπαίνουμε στη δεύτερη φάση τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα ισχύσει σήμερα, για να... αλλά στην επόμενη φάση. Προτείνουμε και βελτιώσεις στην μεταβατική φάση, βελτίωση της εκπροσώπησης και περισσότερη ενοποίηση. Στην πρότασή μας δε αυτό σημαίνει ότι στους τομείς όπου έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου η Ευρωζώνη εκφράσει άποψη, θα πρέπει να είναι ενιαία η εκπροσώπηση. Δεν υπονοούμε τίποτα σχετικά με τις αρμοδιότητες. Μιλούμε για τομείς όπου η Ευρωζώνη έχει, διαθέτει δηλαδή κάποια θέση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στην προσπάθεια αυτή και βεβαίως βασιζόμαστε και στην εργασία που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε ό,τι αφορά την προς τα έξω εκπροσώπηση, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγούν στο να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλούμε για το ποια πολιτική θα υποστηρίξουμε, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι το πώς. Ορισμένοι ευρωβουλευτές συζητούν την ουσία. Εμείς δεν μιλούμε για το ποιες θέσεις πρέπει να στηρίζονται και να προβάλλονται, αλλά πώς θα είναι η ισχυρότερη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλία Σιλβιέτ, δεν είναι και όχι νομοθετική. Δεν προβλέπεται λοιπόν καταρχήν να δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το νόημα της εκθέσεως πρωτοβουλίας είναι να περιλάβουμε σε αυτήν όσα επιθυμούμε εμείς. Η δική μα είναι η πρωτοβουλία, ε, χωρίς τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά βεβαίω καλά κάναμε και την ακούσαμε. Η κυρία Γκούλαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς θεωρώ ότι είναι θέμα ευγένεια να δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή που κάνουν τον κόπο να έρχονται εδώ για ένα θέμα που είναι αρμοδιότητά του. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα όλου. Θα έτσι διαλέξω κάποια στο οποία θα απαντήσω για την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι όντω είναι θέμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οπότε θέλω να πω στον κύριο Τζάνι το εξή. Δεν νομίζω ότι τα δύο παραδείγματα που δώσατε εσείς είναι σωστά. Καταλαβαίνω τι λέτε για το τίλακ και το άλλο. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω πολύ καλά είναι γιατί η μη οργάνωση, προκειμένου να έχουμε ενία φωνή, προστατεύει. Το τίλακ εμφανίστηκε ανεξάρτητα από τους κανόνες που έχουμε υιοθετήσει στα διάφορα ψηφίσματά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι το πώς θα σταθμίσουμε τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με το δημόσιο χρέος, εγώ δεν βλέπω γιατί αν οι αποφάσεις παραμέναν εθνικές, έχουμε καλύτερη προστασία θα ήθελα να το συζητήσουμε γιατί νομίζω ότι ο στόχο μα είναι ο ίδιο. Δεν είναι επιλογή του εισηγητή να πει ότι διαλέγουμε το ένα ή το άλλο επίπεδο. Υπάρχουν συζητήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνε που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των αγορών, το άνοιγμα των συνόρων κτλ. Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι ακόμα και αν θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιε ιδιαιτερότητε, εντάξει, θεμητό, πρέπει να τι υποστηρίζουμε από κοινού. Πάντως, αν δεν τι υποστηρίξουμε από κοινού, οι χώρες δεν έχουν καμία εγγύηση ότι θα μπορέσουν να διατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες αυτές. Οπότε θα ήθελα να το συζητήσουμε από κοινού, μήπω βρούμε κοινό τόπο. Δεν βλέπω πάντως πώς το σύστημα έτσι ω έχει. Άτυπο αποφεύγοντα την πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Να το συζητήσουμε πάντως. Επίσης, σημείωσα και αυτά ε, που είπε μόλι για το συμφωνούμε, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι εκπροσώπηση ενία θέλουμε και σας ευχαριστώ που με οθείτε να είμαι περισσότερο κοινοτική. Ευχαριστώ. Είναι αυτό που είπε και ο Φιλίπ. Ε, πρέπει να το προσέξουμε και εδώ να απαντήσω και στον πρόεδρό μας για το ζήτημα του να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα με την ε, καλή έννοια του όρου, ο, στον FMI για παράδειγμα οι χώρες μέλη ε, συνεισφέρουν επί της ουσίας και αυτό δημιουργεί δικαιώματα στις χώρες μέλη να ξέρουν που πάνε τα χρήματά τους. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι η Τραπεζική Ένωση είναι ένα τομέα περισσότερο ευνοϊκό για να προσπαθούμε να έχουμε ενιαία εκπροσώπηση, ακόμα και αν καταλαβαίνω αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν τελικά συμφωνώ. Η κατεύθυνση πάντως που εμείς θέλουμε να δώσουμε είναι εκείνη της ενιαίας εκπροσώπησης. 20-30 χρόνια, για σκεφτείτε το, πώς είναι δυνατόν θα διατηρήσει τις έδρε που έχει τώρα στα διεθνή φόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 25 χρόνια δεν θα είναι δυνατόν πια αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λες ότι δεν πρέπει να αποδυναμωνόμαστε, να εντοπίσουμε κάποια, κάποιους οργανισμούς. Τώρα για τα λογιστικά πρότυπα, όπως και για το σκιώδες τροπεζικό σύστημα, είναι παραδείγματα αυτά, παρόλο που εδώ η έκθεσή μου δεν εξετάζει την ουσία, αλλά είναι παραδείγματα θεμάτων τα οποία μας βοηθούν να γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες πραγματικότητες. Για την ποικιλομορφία των εποπτικών οργάνων, ναι, με τη δημιουργία της ε, ΕΣΜΑ, της ΙΟΠΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών κτλ είπατε ότι είναι it's a ότι είναι ένα μπέρδεμα. Δεν συμφωνώ ακριβώς, αλλά εντάξει, χρειάζεται περισσότερο εξορθολογισμός. Αυτά. Κατά τα άλλα θα συζητήσουμε στους σκιώδες. Είτε είσαστε σκιώδες, είτε δεν είσαστε. Για παράδειγμα, όποιοι έχουν υποβάλει πολλές τροπολογίες, όπως εσείς, ευχαρίστως να έρθετε. Είμαι στη διάθεση όλων. Και το με το Στην προηγούμενη εντολή υπήρχαν πολλές εκθέσεις με τις οποίες προσπαθούσαμε να είμαστε ενωμένοι εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί κυρίως σε θέματα λογοδοσίας δεν θα εισακουστούμε παρά μόνο να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το πνεύμα, εν πάση περιπτώσει, με το οποίο εξετάζω την έκθεση αυτή. Και χαίρομαι αν κάποιοι από εσά πιστεύουν ότι όντω θα προχωρήσουμε ουσιαστικά. Θα το πετύχουμε αν στηριχθεί ευρέω η έκθεση αυτή, ακόμα και αν κάποιοι έχουν αμφιβολίε, και το αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι έχουν αμφιβολίε για τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά και παρόλο που μπορούν να γίνουν περισσότερε βελτιώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να στηρίξουμε αυτή την έκθεση. Γιατί εγώ εδώ δεν κάνω επιλογέ. Απλώ λέω ότι αν η φωνή τη Ευρώπη μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο, που στηρίζουμε τις ελευθερίες, τη... τα κοινωνικά μοντέλα κτλ. Ο κόσμος θα ήταν χειρότερος αν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε με μία φωνή. Αυτό μόνο λέω. Από εκεί και πέρα όλα τα σχόλια ευπρόσδεκτα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο στη συνάντηση των σκεδών και κατά τα άλλα είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ Σιλβί. Χρονοδιάγραμμα. 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών, Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Θέμα 8. Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών που λέγεται μεταρχικά ΤΙΣΑ και τον λόγο λαμβάνει η συντάκτη της γνωμοδότησης κυρία Αλέσια Μαρία Μόσκα. Σας ευχαριστώ πολύ σύντομα γιατί ε, έχουμε ήδη δει το θέμα. Ε, μάλλον σήμερα είναι μια πρώτη παρατήρηση με μια πρώτη ανάλυση για τις ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Πριν να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες για τις ίδιες τις τροπολογίες, σε σχέση, να πω δύο λόγια σε σχέση με τη 14ο γύρο συζήτησης για το ΤΙΖΑ που έγινε τον Οκτώβριο και γιατί υπήρξαν πευρώδη στα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Ε, πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις δεσμεύσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για τα ε, θέματα μονοπωλίου, θέμα, νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μηχανισμοί αυτορύθμισης. Οι διατάξει σε σχέση με τη διαφάνεια και την εγκρίσεων στον τομέα, το χρηματοπιστωτικό τομέα, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση, συζήτηση και οι συμμετέχοντε συζήτησαν τον κατάλογο ε, για τη δυνατότητα των ε, διασυνοριακών ε, συναλλαγών και υπηρεσιών. Εδώ χρειάστηκε, θεώρησα ότι έπρεπε να σας ενημερώσω γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις. Τώρα, ως προς αυτό, τώρα όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, να πω ότι υποβλήθηκαν 73 τροπολογίες, από τις οποίες 13 υποβλήθηκαν από μένα την ίδια συζητήτρια για να ε, προσθέσω κάποιες αναλύσεις σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότησης που είχα παρουσιάσει νωρίτερα και επίσης υποβλήθηκαν ακόμα 60 τροπολογίες που συζητήθηκαν σε μια πρώτη συνεδρίαση με τους σκιώδεις των ομάδων και άρα ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτές για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να υποβάλουμε κάποιες συνδυαστικές. Τώρα πιο συγκεκριμένα δουλέψαμε με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για μεγάλους τομείς προσανατολισμού. Καταρχήν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις ομάδες, ανάμεσα σε όσους σκοπεύουν να συμπεριλάβουν και πόσους ε, προτίθεται να αποκλείσουν από τις προτώσεις τους τις ίδιες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τη συμφωνία με τη ε, Τίζα ε, Δεύτερον, ε, επίπεδο φιλοδοξίας ε, των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά. Τρίτη ομάδα τροπολογιών αφορά το πεδίο εφαρμογή ε, το ρυθμιστικό κεφαλαίου σε τομέα, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Έπειτα έχουμε τη σύνδεση των διαπραγματεύσεων της ΤΙΖΑ με, τις με τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών και έπειτα ένα άλλο ε, επίπεδο παροχή ε, πληροφοριών διασυνοριακό, για τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιστοιχίας. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τους υποπροηγούμενους και τους ε, σκιώδεις και αυτή η πρώτη σύσκεψη ήταν ε, χρήσιμη για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα κάνουμε πιο αποτελεσματική τη συνεργασία μας. Ως γενική στρατηγική, όπως είχα ήδη τη δυνατότητα να σας πω στην πρώτη παρουσίαση που έκανα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα όριο σε σχέση με αυτές τις τροπολογίες που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής. Αυτό είναι ο γενικότερος προσανατολισμός. Για όλα τα υπόλοιπα έχουν υποβληθεί 10 συμβιβαστικές τροπολογίες που όπως σας έλεγα προσπάθησα να συγκεντρώσω τις προτάσεις των ομάδων Επ' αυτόν εργαζόμαστε. Έχουμε ζητήσει από τις διάφορες ομάδες να μας στείλουν και γραπτός ε, περαιτέρω σχόλια σε σχέση με τα όσα προέκυψαν από την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών και ζητώ και τώρα ακόμα μια φορά όσοι θέλουν να στείλουν ε, τροπολογίες να μας τις στείλουν μέχρι και αύριο έτσι ώστε πριν από την επόμενη συνεδρίαση με τους κοιόδης να μπορέσουμε να έχουμε κείμενα πιο οριστικοποιημένα. Σας έλεγα ότι δουλεύουμε και για την μορφή, για τον τύπο, για όλες τις τροπολογίες προσπαθούμε να μειώσουμε το, τα κείμενα, να τα κάνουμε πιο περιορισμένα και πιο εμπεριστατωμένα, πιο συνεκτικά. Και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτή την γενική συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχόλια, αν υπάρχουν από τους Σκιώδης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ρωμάνα Τόμς. Ευχαριστώ για την... που μας δίνει το λόγο κύριε Πρόεδρε. κυρία Τόσκα εμφανίστηκε ανοιχτή στις ε, προτάσεις μας. Καταλήξαμε σε θετικές συμβαστικές προτάσεις σε λίγο χρονικό διάστημα. Είναι καλές συμβαστικές προτάσεις που γίνονται. Υπάρχουν και ορισμένες προβληματικές, θεωρεί το Λαϊκό Κόμμα. Θα τις πω. Δεν έχουμε βέβαια ακόμα την τελική εκδοχή του κειμένου. Ίσως λοιπόν να δούμε κάποιες αλλαγές. Ας δούμε λοιπόν τις συμβαστικές. Πρώτα, η Α. Σωστή κατεύθυνση και ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία υποστηρίζουμε και την Κομισιόν και τον κλάδο, γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, ρυθμιστικού αρμπιτράζ. Τώρα, η Β. Πρώτο μέρος αντιφάσκει στον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί οι διαπραγματεύσει τα τελευταία δύο χρόνια και αντιφάσκει επίσης στη συμβαστική γάμα, η οποία λέει και σωστά ότι δεν θα πρέπει να ξαναανοίξουν οι συνομιλίε για την διάρθρωση, για τη δομή δηλαδή τη συμφωνία. Άλλο σχόλιο. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο θέμα σχετικό με την εξοεδαφικότητα θηγατρικών ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Ολοδαπή. Μετά, η διατύπωση στη Δέλτα είναι εντάξει. Θα δούμε όμω όταν θα έχουμε το τελικό κείμενο. Συμβαστική ε. Έχει καλώ που λέει ότι ο ΠΟΕ ε, και για τον ΠΟΕ και τι ε, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Όμω υπάρχει μια αντίφαση μετά. Στο σίγμα ΤΑΦ τώρα, στη μαστική σίγμα ΤΑΦ, δηλαδή F, Όμως αυτά τα πράγματα συζητούνται στην ΤΙΣΑ, στο οριζόντιο κεφάλαιο όπου επιγράφεται διαφάνεια. Και εκεί αναφέρεται σε όλους τους τομείς. Εμείς βέβαια συμφωνούμε να παραμείνει εντός. Συμβαστική G, τα θέματα φορολογίας. Έχοντα συζητήσει το θέματα, τα θέματα της ε, φορολογίας με τους συνάδελφους μας της ΙΝΤΑ, που δική τους αρμοδιότητα είναι, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικές, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε και άλλα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να το διατηρήσουμε, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι είναι αρμοδιότητα της ίντα. Για την ε, συμβαστική age η αρχή της είναι ισορροπημένη, αλλά μετά γιατί μιλούμε μετά για financial services που η ροή πρέπει να ε, βελτιωθεί. Γιατί και αντιδρούμε ως Λαϊκό Κόμμα στην αναγκαστική localization. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δηλώσεις για την εντολή και για, την πρόσβαση, και για τις προσφορές πρόσβασης στην αγορά έχουν ήδη καταστεί δημόσιες και μάλιστα και μετά από αίτημα του Λαϊκού Κόμματος. Και τέλος, συμβαστική J, όπως είπα και στην συνάντηση του Σκιωδών, πρόκειται η αντιγραφή από το σχέδιο εκθέσεως της ΙΝΤΑ η οποία μάλιστα τα πήρε από το ψήφισμα για την συμφωνία TTIP. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι μια και δεν έχουμε ακόμα το τελικό έγγραφο, ελπίζω ότι η εισηγήτρια θα δεχθεί να εξετάσει τις, ε, τα σχόλιά μας και θα επανέλθουμε βέβαια. ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο σκιώδης της ECR. Η σκιώδης της ECR, η κυρία Σουίνμπορν. βρίσκομαι τροπολογι... Ε, ε, συμβιβαστικές ε, εδώ και αυτό ήδη είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι στην τελευταία συνεδρίαση. Νομίζω πως ε, εφόσον είμαστε συντονισμένοι θα επηρεάσουμε και την εργασία της Επιτροπής Ίντα, δεν θα αγνοηθούμε. Ωστόσο υπάρχουν τομείς όπου εμείς ε, νομίζω ότι προσθέτουμε αξία στην γνωμοδότηση Υπάρχουν οι διατάξεις GATS που επιτρέπουν την υπογραφή των συμβαλωμένων ε, σε συγκεκριμένες συμβάσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ακυριότητας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τώρα ισχύει αυτό για ένα μικρό ποσοστό των μερών της ΤΙΣΑ. Εγώ υποστηρίζω ότι θα έπρεπε όλα τα μέρη, τα μέρη της ΤΙΣΑ να ε, το συνυπογράψουν αυτό. είναι μια πολιτική προτεραιότητα γιατί η φορολόγηση θα έχει κανονικά τη θέση της σε μια τέτοιου είδους συνθήκη, όμως εγώ υποστηρίζω τους διεθνείς οργανισμούς και τη συμμετοχή μας ε, στις εργασίες αυτές. Εδώ, σε αυτή την έκθεση, ωστόσο, δεν είμαι βέβαια ότι έχουν τη θέση τους. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ, Κέι. Μετ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολη δουλειά. Υπάρχουν κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε με τι οποίε θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αν γίνουν κάποιε αλλαγέ. Με άλλε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Παρά το γεγονό ότι κάποιες τροπολογίες φαίνεται να είναι συμφιλειωτικέ. Η συγκήτρια έχει κάνει όσο μπορούσε περισσότερες προσπάθειες για να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες σοβαρές πολιτικές διαφορές επί του ζητήματος αυτού μεταξύ μας. Και γι' αυτό οι συμβιβασμοί και η συνένεση ακόμα λιγότερο δεν θα επιτευχθούν. Για τις συμβαστικές τροπολογίες ευχαρίστως να σας δώσουμε τις απόψεις μας. Βλέπετε, η κύρια δυσκολία είναι η προσέγγιση για τις εμπορικέ διαπραγματεύσεις της Επιτροπής και γενικά των ε, θεσμικών οργάνων. Και παρόλο που δεν συζητήθηκε αρκετά στην κοινή γνώμη, οι συμφωνίες είναι εκτενέστατες αν μάλιστα λάβετε υπόψη σας και το TTIP και όλες τις άλλες συζητήσεις που έχουν γίνει. Βγαίνουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τις εμπορικές αυτές συμφωνίες όταν προσφέρονται στην κοινή γνώμη. Και βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη ανησυχεί όλους ιδιαίτερους και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Γενικά η κοινωνία για το βαθμό στον οποίο μάλιστα που εκπλήσει από ό,τι φαίνεται τους υπαλλήλου των ε, θεσμικών οργάνων. Ο πληθυσμός που θα επηρεαστεί πάντως από τέτοιες αποφάσεις είναι πολύ μεγάλος όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν όπως έχουν τώρα τα πράγματα δεν θα μπορούσα να στηρίξω την έκθεση αυτή για το ΤΙΖΑ γιατί πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που θα ήθελαν οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες να πάει. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, θετικά κάποιες συμβαστικές προτάσεις έτσι ώστε οι πιο ζημιογόνες ρυθμίσεις να μην περάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ελευθέρωση θα περάσει όσο γίνεται λιγότερο και τα καρτέλ θα έχουν όσο γίνεται λιγότερη δύναμη. Πρόεδρος. Ραϊμόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μόσκα για την έκθεσή της. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα τα σημεία, ιδιαίτερα για τις δημόσιες υπηρεσίες και τη φορολογία. Μάλλον μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποια άλλα στοιχεία κλειδί. Πρώτον, είμαστε κατά και του standstill και του sunset, ε, τις δύο αυτές ρήτρε που αναφέρονται στην έκθεση. Το δεύτερο είναι η προσέγγιση όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι η διατύπωση εδώ ξεπερνάει και τα πλαίσια του TTIP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να μην προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τουλάχιστον έχουμε το κείμενο του TTIP. Που έχουμε για το TTIP δηλαδή. Έπειτα. Δεν μας ικανοποιεί η έγκριση που έχει να κάνει με το ΚΑΤ. Εμείς θέλουμε πιο περιορισμένη διατύπωση για το ΣΥΤΑ για παράδειγμα. Και σας έχουμε στείλει και επιπλέον ιδέες για να πάμε ακόμα πιο μακριά από ότι η διατύπωση για το ΣΥΤΑ. Αυτές είναι οι κύριες ανησυχίες που έχουμε για αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η FTD, ο κύριος Βάλι, ε, Τζάνι, Τζάνι, όχι Βάλι. Μιλώ εξ ονόματος του Βάλη που είναι ο σκιώδης μας εισηγητής. Δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν γιατί συμμετέχει σε μια άλλη συνεδρίαση, σε μια άλλη επιτροπή. Θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω ποια είναι η θέση μας. Δεν υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η θέση που εκφράζει η συγκήτρια στην πλήρη στήριξη της ε, χρηματοπιστωτικής απελευθέρωσης. Όχι μόνο δεν θεωρούμε σκόπιμη αυτή την προσέγγιση, αλλά πιστεύουμε πως αυτή η προσέγγιση ακριβώς δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο η απελευθέρωση η χρηματοπιστωτική από τότε που ξεκίνησε η, η πλήρης εδώ απελευθέρωση, πόσες βλάβες έχει επιφέρει σε ολόκληρη την Ένωση, στην, ε, σε απώλειες θέσεις απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης και πόσο ε, ε, η λυγκιώδη ήταν η πτώση σε φτώχεια ε, και αυτό έχει αποδειχθεί από πολλούς οικονομολόγους ολόκληρο τον κόσμο. Και η πρόταση της εισηγήτριας ε, να καταστεί η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προτεραιότητα της ΤΙΖΑ, να δεσμευτούν κυρίως ε, τα συμβαλόμενα μέρη με ρήτρε ε, standstill, κάτι τέτοιο νομίζουμε πως είναι Αντίθετο με την ε, διαδικασία μεταρρύθμισης του G20 που έχει ξεκινήσει από το 2009 μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας ε, ε, κρίσης και αυτό μπορεί να βλάψει τις συζητήσεις που αφορούν τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχουν ξεκινήσει στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμών. Μιλώ για το τραπεζική, τραπεζικό διαχωρισμό και για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πιστεύουμε λοιπόν πως ε, όλα αυτά είναι αντίθετα με αυτή όλη τη διαδικασία Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, ε, θα ήθελα να τις αποσαφηνίσω. Έχουμε τρία, ε, πέντε βασικά στοιχεία. Καταρχήν ε, θα πρέπει να προστατευτεί το δικαίωμα των κρατών μελών στην ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα, οπότε είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα δικαιώματα των κρατών μελών. Άλλο σημαντικό σημείο είναι ο αποκλεισμό των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από αυτή τη συμφωνία, την ΤΙΖΑ, και εν <coughs> γέννη η καλύτερη προσέγγιση είναι ε, ένα θετικό κατάλογο, δηλαδή να πούμε ποιε είναι συγκεκριμένα οι υπηρεσίε εντό αυτή τη ε, συμφωνία που ε, θα μπορούσαν να λειτουργούν. Πάντω, αποκλείουμε οποιαδήποτε υβριδική προσέγγιση ή αρνητικό κατάλογο. Όσον αφορά τώρα τι ρήτρε που προτείνονται, Οποιαδήποτε ρήτρα standstill ή αναδρομικότητας ε, την απορρίπτουμε και επίσης κάτι ακόμα σημαντικό για μας είναι να υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου εξάντε εκ των προτέρων με διαφανή τρόπο ε, αξιολόγηση από, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε πριν να γίνει οποιοδήποτε βήμα να είναι ως ο αντίκτυπος, οι επιπτώσεις, οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει ένα τέτοιο, μια τέτοιου είδους συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους συναδέλφους που να ζητούν το λόγο, ούτε την Επιτροπή. Οπότε η συγγήτρια να συνοψίσει παρακαλώ. Μάλιστα. Πολύ σύντομα. Προφανές είναι από τις παρεμβάσεις ότι υπάρχει μια ε, απόκληση στο κατά πόσο θέλουμε να συμπεριληφθούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη Συμφωνία ΤΙΖΑ ή όχι. Εδώ θα είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε σύγκληση. Ε, όμως, ε, όπως ήδη υπόθηκε και στη συνεδρίαση των σκιωδών, Καταλαβαίνω τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ομάδες και θα ήθελα λοιπόν παρά αυτή την απόκληση Τουλάχιστον λοιπόν επί άλλων σημείων να μπορούσαμε να δουλέψουμε για να συμφωνήσουμε με όλες τις ανακαλύψουμε μάλλον όλες τις ανησυχίες τις οποίες σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι άμεσα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και γι' αυτό καλό όσους δεν το έχουν κάνει ήδη και το επαναλαμβάνω να μου στείλετε τη σχόλιά σας και τις ενδεχόμενες τροπολογίες μέχρι αύριο ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην οριστική διατύπωση κειμένων για την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να δώσουμε μια επόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση σκιωδών. Να έχουμε έτσι ένα οριστικό κείμενο για να μπορέσουμε να λάβουμε θέση πιο ολοκληρωμένα να προσποθήσουμε να διατηρήσουμε μία γραμμή ευρεία συνένεσης και έτσι να έχουμε και προς την προστιθέμενη αξία που θα δώσουμε στην Επιτροπή Ίντα, την αρμόδια επί της και να τονίσουμε ποιες είναι οι δικές μας ανησυχίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί όπως θυμίζω προσπαθούμε να ασκήσουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει το Κοινοβούλιο να παρέμβει στην ε, διαπραγματευτική διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να εκφράσουμε πιο συγκεκριμένα όσο γίνεται σαφέστερα ποιες είναι οι υποδείξεις που δίνει το Κοινοβούλιο και που θα μπορούσαν πραγματικά να επηρεάσουν τις ε, διαπραγματεύσεις. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διαπραγματεύσεις, σε πάση περιπτώσει εξίσου σημαντικές ε, ε, διαπραγματεύσεις με άλλες που καλούν την προσοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία προβλέπεται εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών την 1η Δεκεμβρίου. Η ΔΕ Επιτροπή ΙΝΤΑ θα ψηφίσει στις 10 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε κάποια ε, χρονική πίεση για να ε, καταθέσουμε τη γνωμοδότησή μας. Και στην Ολομέλεια θα καταλήξουμε τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας σήμερα. Στις 3 το απόγευμα θα συναντηθούμε ξανά για τη συνέχιση των εργασιών μας.